Θα ήθελα να χαιρετήσω εγκαρδιότητα τον Ιωάννη Σαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω ξέρετε, διεξάγουμε τι ακροάσεις με βάση τι τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε για την έγκριση τη Επιτροπή και σύμφωνα με αυτέ τι κατευθυντήριες γραμμέ, το Κοινοβούλιο αξιολογεί του υποψηφίου Επιτρόπου επί τη βάση των γενικών αρμοδιοτήτων του, τη Ευρωπαϊκή του ε, προσήλωση, τη αφοσίωσης, ε, της προσωπικής τους ανεξαρτησίας, τη γνώση του χαρτοφυλακίου του, αλλά και τις ε, δεξιότητες επικοινωνία του. Επίση θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι ο υποψήφιος επίτροπος, κύριος Χάν, είχε απαντήσει γραπτός στις, στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι γραπτές του απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στα μέλη σε όλες τις γλώσσες, καθώς και η δήλωση συμφερόντων. Και όλα αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στους φακέλους των Ευρωβουλευτών. Να σας ενημερώσω επίσης πως η ακρόασή μας θα γίνει με έναν γενικό τρόπο που χρησιμοποιείται για όλες τις ακροάσεις του Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσουμε με 10 λεπτά ανακτήρια εισήγηση του υποψηφίου επιτρόπου και έπειτα έχουμε 2 ώρες και 45 λεπτά για ερωταπαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε ερωτήσεις από όλους τους εκπροσώπους κάθε πολιτικής ομάδας, ε, ε, συγκεκριμένα από τους συντονιστές μας και μετά θα ακολουθήσουμε με τις ερωτήσεις των μελών. Ο κατάλογος που έχουμε επεξεργαστεί, ο κατάλογος αγορετών που, έχουμε, που έχει επεξεργαστεί η γραμματεία ακολουθεί τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση θα βασιστεί στην αρχή του ping-pong, δηλαδή ερώτηση θα ακολουθείται από απάντηση και θα δίνεται ένα λεπτό για κάθε ερώτηση και ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει δύο ε, λεπτά για την απάντησή του. Και αν υπάρχει ε, ε, ανάγκη ή αίτηση για επερώτηση, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ακόμα λεπτό για την επερώτηση και επίση ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει ένα λεπτό για να απαντήσει σε αυτήν. Ε, επίσης θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα της, των επερωτήσεων, των συμπληρωματικών ερωτήσεων θα πρέπει να σχετίζεται με την απάντηση του ε, υποψηφίου επιτρόπου στην πρώτη ερώτηση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον επιπλέον χρόνο για να θίξετε ένα εντελώ νέο θέμα. Οπότε θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ε, επιφυλάσσουμε το δικαιώματο να μην επιτρέψω επερωτήσεις που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. Επίσης, ε, προς ενημέρωσή σας, ε, σα λέω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία catch the eye. Και θέλω να σας ζητήσω να μην ε, υποβάλλετε πολλαπλές ερωτήσεις στο ένα σας λεπτό, γιατί αυτό καθιστά αδύνατο το να απαντήσει ο υποψήφιος επίτροπος σε δύο λεπτά και έπειτα θα είστε δυσαρεστημένοι με την απάντησή του. Λάβετε το λοιπόν υπόψη σας παραμένουμε σε αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συντονιστών κατά τη διάρκεια της ε, τελευταίας του συνεδρίας. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να τηρείτε το χρόνο σας, διότι εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και όπως βλέπετε από τον κατάλογο έχουμε ήδη μία επιπλέον ώρα από την κανονική μας. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η ακρόασή μας μεταδίδεται στο site του Κοινοβουλίου στο ίντερνετ, γι' αυτό να φορέσετε το καλό σας χαμόγελο και να φαίνεστε ωραίοι. Επίσης, θα έχετε πρόσβαση στη ε, πρακτικά. Υπάρχει και ε, θα υπάρξουν και πρακτικά τη ακρόαση. Είναι πολύ ανοιχτό το κοινοβούλιο. Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα τη ακρόαση για οποιοδήποτε θέλει να ρίξει μια ματιά. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιοχάνης, Χαν να μας κάνει τις αναλυτήριες του δηλώσεις σε 10 λεπτά. Έχετε το λόγο. Thank you, Mrs. Chair. Σας ευχαριστώ ε, πολύ, Πρόεδρε. Βέβαια θα κρατήσω τους κανόνες που αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι εδώ παρόν, να ακούσω τις ερωτήσεις σας και να σας ζητήσω να μου επιτρέψετε να είμαι Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική τα επόμενα πέντε χρόνια η περιφερική πολιτική, είμαι σίγουρο ότι οι παρόντες συμφωνούν, είναι μια ιστορία επιτυχίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Ξέρουμε όμως ότι δεν υπάρχουν μόνο φίλοι της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, μέσα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωση. υπάρχουν και ορισμένοι πιο επικριτές, σκεπτικιστές, ε, που πιστεύουν ότι θα πρέπει να ακολουθούν άλλες προσεγγίσεις. Εμείς εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δηλαδή η, περιφερειακή πολιτική είναι μια επιτυχία και ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική για την ε, περιφερειακή πολιτική. Εγώ θα έλεγα υπάρχει μια εναλλακτική, θα ήταν μια ακόμα καλύτερη περιφερειακή πολιτική με μια προσέγγιση ολοκληρωμένη. Και εγώ θα προασπίσω και παρακαλώ με στήριξτε για την πολιτική αυτή γιατί ε, θα πρέπει από κοινού να προασπίσουμε τα συμφέροντα των περιφερειών και των ανθρώπων που κατοικούν στις περιφέρειες αυτές. Η περιφερική πολιτική τα περασμένα χρόνια είχε μια επιτυχή εξέλιξη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς κυρία Χίμπνερ γιατί στο περασμένο σας ρόλο ήσασταν η αρμόδια επίτροπος και ο Σαναφασαβίτσχη στους λίγους μήνες που μπόρεσε να ασκήσει το αξίωμα αυτά συνέχισε στην ίδια οδό. Πρόκειται για ουσιαστικά βήματα από τα οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και τα οποία θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε που είναι ουσιαστικά και αποπαριθούν μια καλή πλατφόρμα για τη μελλοντική εργασία. Καταρχήν πραγματικά η φόρα στρατηγική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Περιφερικής Πολιτικής προς τους ευρωπαϊκούς στόχους. Ξέρω ότι εδώ στο σώμα και εδώ στην αίθουσα δεν υπάρχουν μόνο φίλοι του λεγόμενου earmarking, του καθορισμού ορισμένων κονδυλίων για κάποιες συγκεκριμένες ε, ε, χρήσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση προς όφελος των περιφερειών. Δεύτερον, η πρόθεση και η διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου να προσαρμοστούν οι εκτιμήσεις αυτής, εάν από κοινού καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει πραγματικά εδώ κάτι να κάνουμε. Αυτή η βούληση να υπάρξει δηλαδή η δυνατότητα υπέρβασης κάποιας κοινωνικής αδράνειας θα έλεγα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τέλος επίσης η ιδέα να εξετάσουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα και όχι μόνο να τα εξετάσουμε αλλά και να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Η περιφερειακή πολιτική πάντα εξετάζεται κύριε και κύριοι και ιστορικά εξετάζεται τα τελευταία χρόνια οπωσδήποτε υπό το πρίσμα της ε, ε, ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Αυτό που ήταν χωρισμένο τόσα χρόνια έπρεπε να συνενωθεί πάλι. Νομίζω ότι προχώρησε πάρα πολύ καλά. Και είδαμε ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη σημαίνει οι πιο φτωχές ε, περιοχές και στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια της Ευρώπης να τις έχουμε πάντα κατά νου να εξασφαλίσουμε η οικονομική βάση να υπάρχει για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι σχετικές δομές. Θα πρέπει όλοι να έχουν μια δίκαιη ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κατανομή της ζευμάριας. Τώρα έχουμε με μια νέα πρόκληση, την οποία δεν γνώριζε κανένας μας πριν από κάνα δύο χρόνια. Και πάλι καλείται η περιφερική πολιτική να καταδείξει αποτελέσματα. Όλοι εμείς θα πρέπει να δείξουμε αποτελέσματα. Καμία περιφέρεια στην Ευρώπη δεν έχει μια εγγύηση σε ΣΑΗ. Κάθε περιοχή, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι ίσως σε καλή οικονομική κατάσταση, μπορεί να απειληθεί στο μέλλον. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε σωστές λύσεις, συγκεκριμένες λύσεις για όλες τις περιφέρειες και να τις εφαρμόσουμε όπως πρέπει για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά τους. Και θα ήθελα να σας πω εδώ ξεκάθαρα κυρίε και κύριοι το εξή. Είμαι αντίθετος προς μια επανεθνικοποίηση. Χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχή, μια περιφερειακή πολιτική σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ε, το στόχος δεν είναι ε, ορισμένες ε, περιφέρειες να πάρουν κάποια χρήματα. Δεν θέλουμε, όπως άκουσα να λέει κάποιος, ένα ταμείο φιλανθρωπικό. Όχι, εμείς θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί στις περιφέρειες να δουνε να επενδύουμε σε αυτούς. Και ξέρουμε ότι θα έχουν αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως να εξασφαλίσουμε το ότι υπάρχει καλό. και να το αναπτύξουμε. Και εδώ αναφέρομαι σε τρεις συγκεκριμένους τομείς δράσης. Πρώτος, η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει ξεκάθαρα να τεθεί στην υπηρεσία των κεντρικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγικής 2020. Ανταγωνιστικότητα, η κοινωνία της γνώσης, προστασία του κλίματος και ε, μεταστροφή ε, όσον αφορά την ενέργεια. Αυτό δεν επιτρέπεται να παραμείνουν μόνο κενά λόγια, σλόγγαν, θα πρέπει να ε, τα γεμίσουμε με δράσεις, με αποτελέσματα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με άλλους τομείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρευνα, καινοτομία, παιδεία, περιβάλλον, ε, βιομηχανία, μιμιέψιλον. Ε, όταν το πετύχουμε αυτό τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική προστιθέμενη αξία και να μεγιστοποιήσουμε την πολιτική συνοχής. Και αυτό χωρίς earmarking δεν θα είναι δυνατόν. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και βέβαια επειδή ξέρετε τι έκανα μέχρι στιγμή στην πολιτική μου ζωή δεν θα εκπλαγείτε. Θέλω λέω μια νέα πολιτική για τις πόλεις της Ευρώπης, για τα αστικά κέντρα, γιατί εκεί βρίσκεται η οικονομική, πολιτιστική και ε, κοινωνική ψυχή, αν θέλετε, της Ευρώπης. Τα καυτά σημεία της Ευρώπης και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία εδώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα. Και αν μου δώσετε την εμπιστοσύνη σας, θέλω αμέσως να αρχίσω με βρία διαδικασία διαβούλευσης, ούτω ώστε τα αποτελέσματα να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, το εξής. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια καλή ισορροπία, ισορροπία συγγνώμη, μεταξύ της, ε, του ελέγχου των σφαλμάτων αφενός και της μείωσης όμως του γραφειοκρατικού άχθους αφετέρου. Να πετύχουμε μια ακόμα καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο. Σας το λέω ανοιχτά ότι το ποσοστό σφάλματος που δηλώνει το ελεκτικό συνέδριο για μένα είναι ένα μήνυμα, ένα σήμα προειδοποίησης. Δεν επιτρέπεται να έχουμε καμία ανοχή όσον αφορά την πολέμηση των σφαλμάτων αλλά και ιδίως των απατών. και θα αναλάβω όλα τα μέτρα που μπορώ για να το καταπολεμήσω. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλές καλές δραστηριότητες εδώ τα τελευταία χρόνια και σας λέω ανοιχτά, μια υγιής οικονομική διαχείριση δεν είναι σε αντίθεση με απλούστερες διαδικασίες, με απλούστερους κανόνες. Τα χρειάζομαστε αυτά ούτω ώστε να έχουμε κατανοητούς κανόνες που θα είναι η εγγύηση για μια ελαστιοποίηση του ποσοστού σφάλματος. Και τέλος θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής. Τελειώνοντας κυρίες και πρόεδρε θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά τις ιδέες μου για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ ημών και εμού. Ξέρετε Έχω μεγάλο παρελθόν ως βουλευτής σε μια περιφερειακή βουλή και μετά στη, στο Δημορχείο της ε, Βιέννης. Ξέρω λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα των βουλευτών. Ξέρετε ε, τι σκέφτεται κανένα. Αυτός εκεί στο εκτολιστικό όργανο έχει εκατοντάδες συνεργάτε. συνεργάτες. Εγώ έχω λίγους ξέρω τα προβλήματα αυτά και μπορείτε πραγματικά να είσαστε σίγουροι ότι θα αντιδράσω σε αυτά. Σας χρειάζομαι όμως και όλους γιατί εσείς γνωρίζετε την Ευρώπη, γνωρίζετε τις περιφέρειες, γνωρίζετε τα προβλήματα, τις ανάγκες. Πέστε μου τι χρειάζεται. Θέστε το εδώ επιτάπητος για να κάνουμε κάτι υπέρ των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε αυτό το θαυμάσια ήπειρο. Από κοινού μπορούμε πολλά να πετύχουμε για την Ευρώπη. Προτίθεμαι να το κάνω. Και τώρα προτίθεμαι να απαντήσω στις πολλές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ήταν ιδιαίτερα Συναπαραστατική η δήλωσή σας. Ο κύριος Βανίστελ Ροϊ πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε. Επίτροπε, καλώς ορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω να σας υποβάλω μια ερώτηση που έχει σχέση με το μέλλον μας. Έκανα μια, έκανα μια θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το, μέχρι το 2000, μέχρι το 2020 αλλά ε, φαίνεται να ξεχνάμε ότι θα χρειαστούν για όλα αυτά χρήματα, ένα συγκεκριμένο προπολογισμό. Τι πιστεύετε με αυτή, για αυτήν την αυξανόμενη τάση για την ε, τομεοποίηση, τον κατακαιρματισμό των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Και έπειτα το Ευρωκοινοβούλιο επιθυμούσε ένα λευκό βιβλίο για την εδαφική συνοχή. Υποστηρίζετε αυτή τη νέα προτεραιότητα. Ποια πρόοδο μπορούμε να περιμένουμε σε αυτό το επίπεδο βράχη πρόθεσμα. σα ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο σα. Δύο λεπτά είπατε. Ωραία, θα προσπαθήσω. Βέβαια θα πρέπει από κοινού να καταβάλουμε προσπάθειε. Ούτω ώστε η πολιτική συνοχή να έχει μια, ένα εμφανή ρόλο, εμφανή σημασία και στο γραπτό κείμενο. Το πιο σημαντικό είναι όμως να μπορέσουμε να καταστήσουμε το σεφές ότι μόνο μία προσέγγιση ολοκληρωμένης πολιτικής είναι σε θέση να ε, ικανοποιήσει τις ανάγκες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Αυτή η συζήτηση θα μας κάνει επίσης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να δράσουμε ανάλογα, γιατί και εδώ θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε να υπάρχουν οι επαρκείς πόροι. Και νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον προπολογισμό μέχρι στιγμής είναι μια πολύ καλή βάση για συνομιλίες. Συζήτησα ήδη με διάφορους ενδυνάμει μελλοντικού συναδέλφους ούτως ώστε να προβλέψουμε μια πιο ενδυναμωμένη συνεργασία επί των θεμάτων. Και όσον αφορά την ε, δαφιακή συνοχή και την επικρι... αντιμετώπιση της μέσα στα πλαίσια μιας ευρείας συζήτησης για τις πολιτικές, εγώ είμαι ανοιχτός. Αναρωτιέμαι όμως κατά πόσον ε, μια που θα έχουμε τώρα για λόγους αποτελεσματικότητας στην έκθεση για τη συνοχή ταυτόχρονα προετοιμάζοντας τις εργασίες του μελλοντικού προγράμματος, ε, νομίζω ότι αυτή η Λευκή Βίβλος θα ήταν παραλλήλου μια συμπληρωματική εργασία και θα ήταν καλύτερο να φροντίσουμε τις σκέψεις αυτές να τις εντάξουμε στη μελλοντική, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ. Σημαντική ερώτηση. Ε, ε, Κοιτάξτε, ε, σύνδεση κάνατε με την πέμπτη έκθεση για την συνοχή. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την νομοθετική κατεύθυνση. Ακόμα μια ερώτηση. Μας μας σοκάρισε το, επίσημο, το ανεπίσημο μάλλον έγγραφο για την χρηματοδότηση. Δεν έχουμε ασχοληθεί με το περιεχόμενο, αλλά διαρωτώ με εσείς τι πιστεύετε για αυτή την αναθεώρηση, την ενδιάμεση. Ποια είναι η θέση σας. Και για την περιφερειακή πολιτική ε, ισχύει το κάν το καλό και κουβέντιαζε το κιόλα. Ε, γιατί στην ε, τελευταία περίοδο είχαμε πάνω από 600.000 νέες θέσεις απασχόλησης, πάνω από 100.000 ε, χιλιόμετρα δρόμων. Εκατομμύρια άνθρωποι μπόρεσαν να έχουν καλή τροφοδότηση με καθαρό νερό, να συνδεθούν στα δίκτυα αποβλήτων λιμάτων. Όλο αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να είναι γνωστό τι γίνεται με τα χρήματα που δαπανούνται και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ε, χαιρετίζω και σας καλωσορίζω κυρία Χάνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτηση του Λομπέρ. Είπατε ήδη ότι χρειαζόμαστε ορισμένε αλλαγέ στη μελλοντική ε, πολιτική όσον αφορά τη συνοχή και τις δομές. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε μια πραγματική φιλοκυπαϊκή πολιτική. Εάν ναι, ήταν οι προτεραιότητε για σας. Και μια συμπληρωματική ερώτηση όσον αφορά την ε, δαφική συνοχή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχουμε κανένα ορισμό τι είναι αυτό δεν θα ήταν καλό πριν περάσουμε στη νέα συζήτηση για τη μελλοντική διαρροτική πολιτική να εξετάσουμε το θέμα της εδαφικής αυτής συνοχής για να ξέρουμε τι συζητάμε. Απάντηση. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να σας χαιρετήσω όλους ιδιαίτερος. Ναι, θα πρέπει νομίζω να το συζητήσουμε το θέμα. Οπωσδήποτε δεν έχουμε ακόμα έναν επίσημο ορισμό επιτάπητος. Ούτε και η επιστήμη μπόρεσε να μας βοηθήσει εδώ. Αλλά από αυτό που άκουσα σε πολλές συζητήσεις τους τελευταίους μήνες ε, θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν δίκαιοι όροι σε όλες τις περιφέρειες και αυτό είναι μια πολύ καλή πρόσβαση της ιδέας του πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την ε, περιφερειακή συνοχή, την ε, εδαφική συνοχή, συγγνώμη. Τώρα, όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις, οι σκέψεις αυτές που γίνονται ήδη τώρα για την Ευρώπη 2020, θα πρέπει, εκτός από τη σφαιρική στρατηγική, να είναι ο στόχος μας, να υποστηρίξουμε δηλαδή την κοινωνία της γνώσης, να αναπτύξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά μην αφήσουμε και κατά νου τα θέματα της υποδομής. Και σας το λέω ξεκάθαρα, κοιτώντα τι γίνεται εν ώψη της κρίσης σε όλες τις χώρες για την ενδυνάμωση της ε, έρευνας και της ανάπτυξης και κοιτάω μετά όμως τους προϋπολογισμούς τους σχετικούς που βλέπω ότι έχουν περικοπεί σημερικά. Βλέπω ακριβώς εδώ το έργο της Ένωσης να είναι παραδειγματική, να επιμείνει εδώ να υπάρχουν συνέργειες. Εδώ καλύπτε, καλείται συγγνώμη, η Ένωση να δώσει το καλό παράδειγμα και εν αντιθέσει προς την αρχή της επικουρικότητας να αναλάβει η Ένωση την ευθύνη, ούτως ώστε και στην κρίση να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, μια που ξέρουμε πόσο κατεπηγόντως χρειαζόμαστε την έρευνα και την ανάπτυξη αυτή για να βγούμε πιο ενδυναμωμένοι από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ, Κωνσάντσα, στην ερώτηση. Με μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που είπατε. Έχουμε και εμείς παρόμοιες ιδέες. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια ακόμα για το πώς θα μπορέσετε να παρασύρετε μαζί σας τους πολίτες. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή, να περάσουμε σε μια κοινωνική συνοχή. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι μόνο με μια ολοκληρωμένη πολιτική μπορούμε να κινήσουμε κάτι. Χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένα άτομα ήδη στα παιδιά, στους νέους, ούτω ώστε να δημιουργήσω το απαραίτητο δυναμικό για τα πανεπιστήμια. Και χρειαζόμαι από την άλλη μεριά τους επιχειρηματίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και χρειαζόμαστε την αγορά και τους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους πόρους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη πολιτική συνολικά και εδώ συγκεκριμένα να έχουμε πάντα κατά νου τα συγκεκριμένα προβλήματα κάθε περιοχής που μπορεί να δώσει τις συγκεκριμένες λύσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή τις γνώσεις ε, των περιφερειών από κάτω προς τα πάνω για να μπορέσουμε να συναρτήσουμε την πολιτική μας και αυτό θεωρώ μια προχωρημένη, προηγμένη, επιτυχή περιφερική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ραμόνα Νικόλα Μανέσκου. Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χάνα, τον υποψήφιο επίτροπο και ελπίζω πως θα συναντιόμαστε τακτικά και εσείς κύριε Χάνα θα είστε στη θέση του επιτρόπου. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά στην έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής που εστιάζει στην δημιουργικότητα και την καινοτομία ως δύο μέσα που μπορούν να ε, σώσουν ε, νωρίτερα και σωστότερα τα κάτι μέλη από την οικονομική κρίση. Επίτροπε, εσείς πιστεύετε πως η ανάπτυξη των ε, τοπικών ε, ταλέντων και η ανοχή όπως περιγράφονται σε αυτήν την έκθεση προόδου είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ε, εξέλθει της κρίσης. Σας ευχαριστώ. Ένας τομέας είναι αυτός και οπωσδήποτε όχι ο λιγότερο σημαντικός αλλά καμιά φορά υπάρχουν προσπάθειες να μειωθεί κάτι. Ε, ε, θα πρέπει να έχουμε τη σωστή προσέγγιση. Η δύναμη της Ευρώπης όμως ε, μας δίνει δυνατότητα ε, μιας πολυμορφίας και άμα συγκρίνω εγώ την Ευρώπη με άλλες περιφέρειες του κόσμου που δεν έχει την πολυμορφία αυτή βλέπουμε ότι δεν έχουμε τόσο υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας όπως υπάρχει εδώ. Η πολυμορφία είναι στη βάση της ε, δημιουργικότητας. Το ότι η Ευρώπη είχε μια ιστορία επιτυχίας εδώ και πολλούς αιώνες και θα έχει πάλι δεν ήμασταν τόσο πολύ σχετικά στο παρελθόν, ούτε είμαστε και τώρα, αλλά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την πολυμορφία μας αυτή. Και γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε ακριβώς τη δυνατότητα καινοτομία που έχουμε, να το καλλιεργήσουμε αυτό στα παιδιά, στα νηπιαγωγεία ήδη. Αυτές οι συζητήσεις πώς οργανώνουμε, τι κάνουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μέχρι 6 χρονών πώς θα μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν κάποιο ενθουσιασμό για αυτό που κάνουν. Γι' αυτό είναι πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και είμαι πεπισμένος ότι η συνάδελφος στον τομέα της παιδείας θα έχει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες και σας καλώ να κάνουμε κάτι από κοινού. Mulțumesc, domnule Hans.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 ναι, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Ελπίζω πως θα ληφθούν απόψη και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις πολιτικές συνοχές. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο έγγραφο της Επιτροπής για τη Μελλοντική Στρατηγική για Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Θα πρέπει να αναφέρουμε στις τοπικές αρχές πώς πιστεύετε πως όλα αυτά θα εφαρμοστούν τοπικά και περιφερειακά χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και τι σκοπεύετε για να κάνετε ως προς αυτό. Μα γι' αυτό αναφέρθηκα αυτό το και ειδικό και βάρος για τις αστικές περιοχές. Θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και άμα το κάνουμε θα έχουμε και τα σχετικά αποτελέσματα. Είχε πει 150% πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε τους τοπικούς παίκτες, αλλά χρειαζόμαστε και την κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο να μπορέσουμε να κινήσουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν θέλουμε μόνο πολιτικά, διοικητικά να ε, κάνουμε κάτι, αλλά θέλουμε να οργανώσουμε πολλά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά όχι πολύ εμφανώς. Και αυτές οι οργανώσεις θα πρέπει να τις ενδυναμώσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια μιας σφαιρικής στρατηγικής να εφαρμόσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα και να τα εντάξουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστώ, κύριε Φρανσουά Αλφόνζη. Εδώ βρίσκομαι, εδώ βρίσκομαι, κύριε Επίτροπε. Καλώς ορίσατε. Η ομάδα μας θα ήθελα να σας υποβάλει τρεις ερωτήσεις. Ε, Είστε αυτή τη στιγμή κατά της κρατικοποίησης ε, των ε, περιφερειακών πολιτικών, γι' αυτό χαιρόμαστε. Η απάντησή σα είναι πολύ πιο σταθερή και ξεκάθαρη από τα όσα είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. ω επίτροπο μιας χώρα με έντονη αποκέντρωση, θα ήθελα να αυξηθεί ο ρόλος των περιφερειών ε, στη μελλοντική ανάπτυξη και αυτό σε χώρες που έχουν πολύ πιο κεντρική ε, διακυβέρνηση. Έπειτα, πολιτικές και προτεραιότητες ε, της Ένωσης, αλλά θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται και από, ε, και από δημοσιονομική προτεραιότητα. Εδώ πώς μπορείτε να μας καθησυχάσετε. Και έπειτα, στην Επιτροπή μας θα θέλαμε να, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να μπλέκεται όλο ένα και, πιο, και περισσότερο σε, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασία και με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς αυτό. Καταρχήν, αυτό ένα τμήμα τη Ευρωπαϊκή Παραγωγικότητα και τη συνθήκη δεν μου αρμόζει εμένα να τροποποιήσω εθνικές δομές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τις περιφέρειες, να ενδυναμώσουμε αυτή την συνεργασία και όχι μόνο με τις περιφέρειες, αλλά και με την, τους τοπικούς φορείς. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ήδη αναφέρθηκα στον προπολογισμό. Έχουμε σήμερα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό του προπολογισμού. Θα είναι φιλόδοξη η προσπάθεια να το διατηρήσουμε και γι' αυτό θα χρειάζεται συνεχώς να διευκρινίσουμε τι μπορεί να αποφέρει η περιφερειακή πολιτική, πού είναι η προσθεθόμενη αξία της περιφερειακής πολιτικής σε σχέση με μια καθαρά τομιακή προσέγγιση. Ακριβώς εάν τώρα στη νέα συνθήκη θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι για την απεικορικότητα και το έχουμε γράψει αυτό, τότε η περιφερική πολιτική ε, θα πρέπει πραγματικά να ασκήσει αυτή την επικουρικότητα. Και γι' αυτό νομίζω έχουμε πολλές δυνατότητες δράσης, πολλές εναλλακτικέ. Και το τελευταίο σημείο τι ήτανε? ο τρόπος με τον οποίο η δική μας Επιτροπή και γενικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμπλακεί. Ναι, συγγνώμη, πώς το ξέχασα. Πω, πω, πω. Ειλικρινά, με πολλές προσωπικές αλλά και επίσημες επαφές. Και θα ήθελα να σας καλέσω για κάτι τέτοιο. Όσο μου επιτρέπει το χρονοδιάγραμμά μου, να έχουμε μια πολιτική της ανοιχτής πόρτας θα έλεγα. Εγώ δεν είμαι εκείνος που επιμένει μόνο στις επίσημες επαφές όπως έχουν συμφωνηθεί. Πολλά νομίζω μπορούν να ε, συζητηθούν και να επιληθούν σε ανεπίσημες επαφές. Και θα ήθελα να σας καλέσω και εσάς από πλευρά σας να αναλάβετε πρωτοβουλίες, να τις συζητήσουμε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε αλλά το Κοινοβούλιο, το είπα και εισαγωγικά, για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος, γιατί ακριβώς εσείς εκπροσωπείτε τις περιφέρειες Ευρώπης, έχετε τις γνώσεις, τις πολύμορφες, της κατάστασης επιτόπου. Γι' αυτό σας χρειάζομαι και θα μπορούσατε σε μένα να βρείτε έναν ε, βάσιμο συνομιλητή που θα μπορούσε έγκαιρα να σας ακούσει και σας παρακαλώ να μου παρουσιάσετε έγκαιρα τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Ε, γι' αυτό επέτρεψα και στον Επίτροπο να μιλήσει λίγο περισσότερο. Τώρα περνάμε στον κύριο Όλτβιχ Βλάσακα. Συγχαρητήρια κύριε Χάν για το χαρτοφυλάκιό σας. Όπως θυμάμαι από τον δήλωση του κυρίου Μπαρόζο, είναι μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές και ελπίζω και αναμένουμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι θα συνεχίσετε το έργο των προκατόχων σας, όπως η κυρία Χούμπνερ και ο κύριος Σαμέτσκι. Στις γραπτές σας απαντήσεις ε, σημειώνουμε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, θεωρείται πολύ σημαντική. Η εξωτερική ανταγωνιστικότητα αναμφίβολα είναι ένα σημαντικός στόχος για τις κοινοτικές πολιτικές που δικαιολογεί την ύπαρξη τη ίδια τη Ένωση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντοτε το έργο της πολιτική συνοχής και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό να προωθήσει δηλαδή την εσωτερική συνοχή της Ένωση, ε, προωθώντα την εσωτερική ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός περιφερειών και πόλεων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέες επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών. Αυτό ε, για να, μπορέσει να μπορέσουν να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ελεύθερη δηλαδή κυκλοφορία και την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Χάν θέλω να σας ρωτήσω εάν θα μπορέσετε εσείς να σχηματίσετε τη μελλοντική γενεά της ε, πολιτικής συνοχής να την ε, δρομολογήσετε στην αρχική της πορεία ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες και να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την καλύτερη παραγωγικότητα και την ευημερία εάν βλέπετε πως ε, θεωρείτε μάλλον ότι είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα η εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την επόμενη γενεά της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Πιθανότατα δεν θα δοθεί εδώ χρόνος για επερώτηση. Κύριε Χάν. <clears throat> Ναι. Και τούτον πει και το άλλο μία φιέτο θα έλεγα. Η θα πρέπει για τις στοχότερες περιοχές να βρεθούν δυνατότητες και θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε σε αυτό, να καλύψουν τα κενά. Από την άλλη μεριά και οι πλουσιότερες περιοχές βέβαια δεν θα παραμείνουν στάσιμες. Όποιος παραμένει στάσιμος τον ξεπερνάνε τα γεγονότα. Και γι' αυτό θα πρέπει οι λιγότερο καλά ανεπτυγμένε περιφέρειες να έχουν μια καλύτερη δυνατότητα δυνατοτήτων, γι' αυτό τους δίνουμε και περισσότερους πόρους για να καλύψουν το κενό, την καθυστέρηση που έχουν. Και γι' αυτό θα πρέπει αφενός να ε, επενδύσουμε στους κλασικούς τομείς, όπως παραδείγματος κάνει ανάψυξη των υποδομών, υποδομών, να βελτιώσουμε το περιβάλλον, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να κάνουμε και κάτι για την ανάπτυξη κοινωνίας της γνώσης και επίσης να κάνουμε κάτι για τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και να αναπτύξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την ε, την ένταση της ε, δέσμευσης που θα έχουμε και ταυτόχρονα θα πρέπει βέβαια να βοηθήσουμε τις περιφέρειες να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αλληλοστηριχθούν ούτω ώστε να πετύχουν μια σφαιρική κοινή ανάπτυξη. Αυτά είναι τα κυρία σημεία προς τα οποία θα θέλουμε να κινηθούμε. Εγώ σας προεδοποιώ γιατί αυτό θα έχει πάλι αντίκτυπο στην πολιτική μας εάν δεν πρέπει να περιοριστούμε σε ένα πράγμα. Ναι, έχουμε τα κεντρικά μας σημεία και μέσα στα πλαίσια αυτών των κεντρικών σημείων υπάρχουν πολλές δυνατότητες μεμονωμένης προσωπικής πραγματοποίησης συγκεκριμένη της ανάγκης κάθε ε, ε, περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε υπερώτηση, ελπίζω όχι. Α, μισό λεπτό. Πάρα πολύ σύντομη θα είναι η υπερώτηση. Είστε έτοιμος. πώς να το πω, για να καταφύγετε σε αυτές τις μεταβατικές περιφέρειες. Ναι, βέβαια. Οι λεγόμενες ε, ε, μεταβατικές ε, περιφέρειες, τις οποίες θα παρουσιαστούν τις επόμενα χρόνια, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί υπάρχει δηλαδή μια περιφέρεια η οποία σήμερα στο phasing in και στο phasing out ε, ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες όμως που έχουν περίπου το ίδιο επίπεδο αλλά δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, δεν έχουν την ίδια αξιολόγηση. και θα πρέπει να έχουμε πιο απλό σύστημα γιατί αυτές τις πολλές δομές του phasing in και phasing out θα πρέπει να τις μειώσουμε την επόμενη φορά, να τις ενοποιήσουμε και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον περιφέρειες οι οποίες σήμερα βρίσκεται ε, μεταξύ του κατοφλίου 75% και του κατοφλίου 90% αν θα πρέπει αυτές να τις λάβουμε ξεχωριστά υπόψη ή όχι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λιώρα. Κύριε Επιτροπή. Και για την αποτελή περιφέρεια, Ζόρες, ε, Κανάρια, Γουαδελούπη, Μαρτινίκη, Ρενιόν και αυτά είναι στο χαρτοφυλακείο σα. Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία θα υποβάλουν ένα μνημόνιο την επόμενη χρονιά στο, στην Επιτροπή ε, γιατί κάτι το οποίο έχει σχέση με την πρόκληση του 2020. Μπορείτε να μας πείτε εν ώψη αυτής της κίνησης εσείς πώς λογαριάζετε ε, να προχωρήσετε για την απότερη περιφέρεια της κοινότητας σε σχέση με όσο ορίζει η Συνήθεια της Λισαβόνας. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ούτως ώστε η να μπορέσει η, ομάδα εντερσερβής η ε, διαϋπηρεσιακή να μπορέσει να προχωρήσει και κάθε φορά ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της επιτόπου να μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται. Θεωρώ ότι αυτές οι περιφέρειες, οι λεγόμενες outermost regions, αποτελούν ιδιαίτερο πλούτο της Ευρώπης. Αξίζουν τις προσοχές μας και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι οπωσδήποτε θα τα λάβω αυτά όλα υπόψη μέσα στα πλαίσια των μοδιοτήτων. Εδώ και αρκετό καιρό, δεν ξέρω ακριβώς από πότε, στην Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής υπάρχει και αυτή η ομάδα που λέγεται Outermost και που είναι ο συνομιλητής για τις περιφέρειες αυτές για το σύνολο της Επιτροπής. Έχουμε δηλαδή ε, μία διαχείριση με, με μία μοναδική θηρίδα, one-stop shop. από την άλλη μεριά μας προσφέρουν οι περιφέρειες αυτές μία θαυμάσια ευκαιρία να αναπτύξουμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές αξίες με μια καλή πολιτική γυπνίασης και που οι περιφέρειες μας αποτελούν μια βάση. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Μια που δεν έχουμε περώτηση, πάμε τώρα στον κύριο Μπάφτον. Μπάφτον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Χάν. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω με κάτι με το οποίο και εσείς αρχίσατε. Όταν είπατε ότι ορισμένοι είναι επιφυλακτικοί, σκεπτικιστές στην αίθουσα αυτή και μεταξύ αυτών μπορεί να συγκαταλέγετε και εμένα γιατί Κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό γίνει ελπίζω να είναι όχι το αποτέλεσμα και να μπορούμε να χάσουμε τις δικές μας πολιτικές. Εγώ έχουμε από την Ουαλία και ξέρετε ότι έχουμε πάρει χρηματοδότηση ε, και θα την παίρνουμε μέχρι το 2013. Ε, και είναι αυτά τα χρήματα που έχουμε εισφέρει, <clears throat> βέβαια, και τα οποία ε, τώρα τα παίρνουμε πίσω. Οπότε, για πέστε μου τα εξής. Όταν ε, τερματιστεί αυτή η περίοδος του 2013, τι εγγύσει μπορεί να μα δώσετε ότι κάποιε χώρε όπω η Ουαλία πρόκειται να, να, να, να έχουν κάποια ρύθμιση αξιοπρεπή μεταβατικού είδου. Γιατί αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι όσο μεγαλώνει η Ευρωπαϊκή ΕΕ, η ε ε και έχουμε τέτοιες διευρύνσεις, μπορούμε να πάρουμε και την Ισλανδία του χρόνου ή την Τουρκία, οι χώρες οι οποίες μπαίνουν τώρα είναι φτωχές χώρες και φοβάμαι ότι εμείς θα βγούμε Χαμένη. Παρά το ότι είμαστε πλούσια χώρα θα βρούμε χαμένοι γιατί ακριβώ μπουν αυτές οι χώρε. και θεωρώ ότι θα μας ρίξετε όσον αυτή τη χρηματοδότηση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υπάρξει κάποια διαβεβαίωση σχετικά με αυτή μας την ανησυχία. Κύριε Βαφν, ήδη όταν απάντησα στον κύριο Βλάντα και είχα πει ότι οπωσδήποτε αναγνωρίζω την αναγκαιότητα όπως και τώρα και στο μέλλον να φροντίσουμε εκείνες τις περιοχές οι οποίες ευτυχώς λόγω της επιτυχούς περιφερικής πολιτικής βελτιώνουν το καθεστώς τους χωρίς να έχουν φτάσει όμως εκεί που θα πρέπει να φτάσουν αν θέλετε σε αυτές τις περιπτώσεις λέγω ότι θα έχουμε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις και αυτό θα ισχύσει οπωσδήποτε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Βέβαια πάντα υπό τη σκοπιά ότι εμείς από κοινού θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια απλούστευση των κανόνων. Ταυτόχρονα όμως θα αναγνωρίσουμε ότι εκείνες οι περιφέρειες οι οποίες εντάσσονται εκεί λόγω των τιμών τους, αλλά που ότι ποτέ δεν ήταν σε τόσο κακή η κατάσταση όσε άλλε και δεν υπέπιπταν σε αυτή τη μεταβατική διάταξη, θα πρέπει πραγματικά να ενισχυθούν. Αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουν στις λεπτομέρειές του, αλλά νομίζω ότι η Ολία ωφελήθηκε στο παρελθόν από το ότι ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά από πέντε χρόνια, κύριε Βάφτεν, ίσως και εσείς θα είσαστε πεπισμένος Ευρωπαίος. Άμα δείτε ποιες είναι οι, δυσκ... δυνατότητες που ανοίγουν για την Ουαλία λόγω του ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ να το πετύχω από τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ για τόσο είπατε κύριε Αλλά νομίζω ότι Το θέμα είναι κατά πόσο θα χρειάζεται να συνεργαστούμε για να ρυθμιστούν λεπτομέρειε πάνω στι οποίε δεν είπατε τίποτα. Γιατί πολύ ωραία τα πανηγύρια για τι διευρύνσει, αλλά εμεί είμαστε πλούσια χώρα, θα χρειαζόμαστε πίσω τα λεφτά. Ε, δεν έχει λεφτά η ε, ΕΕ. Ε, ε. Ίσως έχουμε κάπως διαφορετικές απόψεις, αλλά καλό είναι αυτό. Και αυτό νομίζω είναι το ωραίο της Ευρώπης, ότι υπάρχει αυτή η πολυμορφία. Είμαι παρόλα αυτά πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Την είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν και θα την έχουμε και στο μέλλον. Επ' τη είμαι πεπισμένος ότι θα τα ωφεληθεί και η Ουαλία. Τις λεπτομέρειες θα τις εξετάσουμε. Από κοινού θα συνεργαστούμε γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ότι όχι μόνο εισφέρει χρηματικά η Ουαλία, αλλά μας δίνεται τρομερή έμπνευση όσον αφορά γενικότερα την οικονομική διαχείριση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική. Επομένω, σα χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη και στην περιφερειακή πολιτική. Και τώρα, για να δούμε τι γίνεται με τα καθέκα των μέλη τη Επιτροπή. Έχετε λιγότερο χρόνο τώρα, ο, ο καθένα. Παρακαλώ, εγώ μόνο ερωτήσει και τις παρατηρήσει και τα σχόλια αργότερα. Κύριε Πίπερ. Πίσω σας κάθομαι, κύριε υποψήφια επιτροπέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε ότι δεν πέτυχε ακόμα η επιστήμη να ορίσει την ε, γεωγραφική συνοχή. Εγώ θεωρώ ότι κανένα δεν το καταλαβαίνει στην ε, πατρίδα μου και το 90% των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο επίση δεν μπορούν να το ορίσουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητάμε περισσότερο αφρική πολιτική ε, υποστήριξη κλπ. Και, και όχι κάποιου όρου που δεν καταλαβαίνει κανένα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην υιοθέτηση τη περιφερειακή πολιτική. Συζητάμε για χρήματα αυτή τη στιγμή. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που πετύχαμε. Αλλά αυτό που μα έλειψε τα τελευταία χρόνια από την Κομισιό είναι να είναι ο συνήγορο των περιφερειών. Υπάρχει μια διαδικασία επιπερεβάση ε, στην ε, Κομισιόν κατά της Γερμανίας ε, γιατί υπάρχουν κάποιες χωροταξικές ε, διατάξεις που ισχύουν. Ποιο προσπίζει τη χωροταξία εδώ, δεν μου απάντησε κανένας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, της Ευρώπης για κάθε λεπτομέρεια σε όλη την περιφέρεια. Εσείς μέχρι πού θεωρείτε ότι φτάνει η αρμοδιότητά σας, κατά πόσον είσαστε συνήγορος των περιφερειών και των περιφερειακών συμφερόντων. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος και έτσι έχω μια διαφορετική εικόνα. Θα θεωρούσα, αν με υποστηρίξετε, ε, ότι είμαι ο πατέρας των περιφερειών. Σοβαρά. Ο κάθε πατέρας έχει συμφέρον τα παιδιά του να αναπτυχθούν καλά, κάνει κάθε προσπάθεια για να έχουν μια καλή ανάπτυξη και να βρίσκονται σε καλύτερη θέση. Καμιά φορά πρέπει να είναι και αυστηρό κανένα όμω. Και να πει εδώ έχουμε φτάσει στα όρια. Ω εδώ και μην παρέκει. Μια που οι αποφάσει στην Επιτροπή είναι βέβαια συλλογικέ, εγώ με την ομάδα μου θα παρατηρήσω, συνεχώς θα παρατηρώ προσεκτικά. Όλες οι ατάξεις που έχουν οι και τοπικές επιπτώσεις χωρίς να είναι της δικής μου άμεσα αρμοδιότητες. Υπάρχει αυτή η ιδέα που κυκλοφορεί και μέχρι να μόνος προς μπορώ να τον κατανοήσω ότι μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης των επιπτώσεων θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες περιφερειακές πτυχές που θα εξετάζονται. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε πιο ανεπίσημη μορφή συνεργασίας, ούτως ώστε εκεί που αναφέρονται περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, να μπορούν αυτές να ληφθούν ανάλογα υπόψη. Και αν δεν ληφθούν επαρκώς υπόψη, να ζητήσουμε να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Μπορώ να σας πω όμως ότι θα προσπαθήσω πάση θυσία να το προωθήσω αυτό. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση όσον αφορά την υιοθέτηση της περιφερικής πολιτικής. Πώς διαβλέπετε εσείς την συνεργασία μεταξύ της ε, διαρθρωτικής ενίσχυσης και της πολιτικής για την υπεθρό που χρηματοδοτείται από την ε, αγροτική πλευρά. Καμιά φορά χρειαζόμαστε παράλληλη χρηματοδότηση, γιατί η χρηματοδότηση γίνεται από διάφορα ταμεία. Μήπως θα μπορούσαμε να τα συνενώσουμε αυτά. Απάντηση. Στην, περιφερική, ε, πολιτική βλέπουν τα πράγματα βέβαια διαφορετικά. Θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά ομολογώ ότι η δική μου προσέγγιση θα είναι μαζί με τους συναδέλφους να πετύχω καλύτερη συνεννόηση, ένα διάλογο Ξέρω ότι υπάρχουν βέβαια κάποιες δυνατότητες και κάποιος κίνδυνος επικαλύψεων και έτσι ορισμένα πράγματα μένουν εκτός, αν θέλετε, της εξέθεσης και είμαι πεπισμένος με καλύτερη συνεννόηση, με καλύτερο συντονισμό των δύο ταμείων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν δυνατότητες ακόμα και εν ώψη μιας ε, καλύτερης ενερμόνησης των κανόνων που εφαρμόζονται. και έτσι να βελτιωθεί η εκμετάλλευση για τον τελικό χρήστη. Και αν υπάρχει καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των δύο ταμείων, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα και θα πρέπει αυτός να είναι ο στόχος μας και θα είναι μία από τις πρώτες μου προσεγγίσεις της εργασίας μου. Κύριος ε, Σταυρακάκης, τώρα κύριε Επίτροπε, εδώ πίσω σας στο έδρανο. Αγαπητέ κύριε υποψήφια επίτροπε. Βεβαίω, κοίτα, θα διαφωνούσατε για το ότι η Ευρώπη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι κοινωνικέ, οικονομικέ και περιβαλλοντικέ προκλήσει, θα πρέπει να συνεχίσει την υποστήριξη τη καινοτομία και τη έρευνα σε κάθε επίπεδο ευρωπαϊκό και διεθνό. Παρ' όλα αυτά όμω, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ενισότητε μεταξύ των περιφερειών. όσον αφορά τις ε, δαπάνες και υπάρχουν κάποιοι, κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που ξεχωρίζουν. Όμως μιλάμε τώρα για κοινέ πολιτικές και θα πρέπει καμία περιφέρεια να χάσει το τρένο. Οπότε με δεδομένο το παρελθόν σας ως ε, Υπουργού Έρευνας και, και, και, Επιστημών τι θα κάνετε τούτος ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό και να μπορέσουν ε, οι επιτροπές που έχουν, οι που έχουν μείνει πίσω να φτάσουν αυτές που προηγούνται σε αυτούς τους τομείς. Κύριε Σταυρακάκη, δύο λεπτά έχω δυστυχώς για να σας πω ε, ό,τι έχω να σας πω. Εγώ θα μπορούσα δύο ώρες να σας μιλάω και να σας αναπτύξω τι μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς αυτή είναι η αλλαγή μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για την έρευνα και του Επιτρόπου για την Περιφέρεια. Γιατί η Ρευνά, για να πούμε ειλικρινά, δεν ενδιαφέρεται πού εκφράζεται η τελειότητά της. Περιφερειακά δηλαδή δεν ενδιαφέρει, ενώ η περιφερειακή πολιτική έχει συμφέρον οι γνώσεις και εξ αυτού οι δυνατότητες να διαχύνονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη κατά δυνατόν. Είναι διαφορετικά κέντρα βάρους βέβαια. Και γι' αυτό εγώ ως Υπουργός Επιστημών είχα μια πλατφόρμα με τους υπουργούς ε, των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης γιατί θέλαμε να αποφύγουμε να υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρώπης ένα λεγόμενο brain drain, μια απορρόφηση εγκεφάλων και θα πρέπει να έχουμε μια κυκλοφορία εγκεφάλων αν θέλετε. Αυτό που δεν θέλουμε και που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι μια συγκέντρωση της ε, επιστήμης, της έρευνας κορυφής σε όλα συγκεκριμένα σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι θα απορροφηθούν εκεί όλοι οι καλύτεροι εγκέφαλοι της Ευρώπης. Θέλουμε να έχουμε πολλές ιδέες, παραδείγματο χάρη ε, προγράμματα υποδομής επιστήμων με δορυφοριακά προγράμματα όπως λέμε. Ο χρόνος που έχω εδώ τώρα να σας μιλήσω λίγη, αλλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλές ώρες και αν θέλουμε θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει η κατανομή να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σαν βάση. Τα πανεπιστήμια είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων έρευνας που θα εφαρμοστούν μετά και στον επιχειρησιακό τομέα. Thank you, Commissioner. You have just... Ευχαριστούμε. Υποσχεθήκατε μόλι τώρα. Εάν όλα πάνε καλά, να έρθετε για να μα μιλήσετε για καινοτομία και έρευνα και για το τι μπορούμε από εκείνο να κάνουμε. Ο Γιάννη Μπρεζίνο. Κύριε Χάνη από ό,τι φαίνεται εύκολη είναι η ερώτησή μου. Για πες μας. Σε σχέση με το όσα για την επόμενη ε, περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής, εσείς θα σεβαστείτε τις ιδιομορφίες των, του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, τι θα κάνετε το, με το Κοινωνικό Ταμείο, θα, διαχωριστεί από τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό, μόνο αυτό. Ich weiß ja, dass die einfachen die, die schwierigsten sind oder die, die äh, ε, οι απλέ ερωτήσει είναι οι πιο δύσκολε και οι πιο ενδιαφέρουσε πολιτικά. Δηλαδή και εδώ ολοκληρώνει το κύκλο. Ολοκληρωμένη περιφερική πολιτική έχει και το Περιφερικό Ταμείο είναι ένα κεντρικό σημείο των, της κοινωνικής ε, συνοχής και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρχει στο μέλλον καμία τροποποίηση των δομών όσον αφορά το κύριο του έργο των διαρθρωτικών ταμείων και μη συνεχής. Όσον αφορά βέβαια την απόδοση θα πρέπει, είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχει συνεργασία. Καταρχήν όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε καθόλου από τις αρχές που διέπουν τα ταμεία αυτά. Evgeny Kirillov. Thank you. Where are Madam Chair. Here, to the left. Ο Ευγέννη Κυρίλοφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφι, Επίτροπε. Υπάρχουν ε, δύο περίπλοκες και βαριές διαδικασίε για τη χρήση των διαθωτικών ταμείων και έχουν επικριθεί γενικώ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τους δικαιούχους. Είναι πρόβλημα αυτό. Και μάλιστα πρόσφατα άκουσα ότι είναι πρόβλημα και για τη δική σας χώρα, που δεν είναι καινούριο νέο κράτος μέλος. Ορισμένοι όταν ακούνε για τα διευθυντικά ταμεία και τα χρήματα από αυτά λένε «Ε, καλύτερα να πάμε στην τράπεζα να ζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι είδου μέτρα προβλέπετε για να ξεκινήσουν απλοποιήσεις και την απλοποίηση τη θεωρείται ως συνεχιζόμενη διαδικασία, γιατί προφανώς μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας θα ολοκληρωθεί η εργασία μας ως προς αυτό το τομέα. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και την επόμενη περίοδο. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν από αυτό. Ναι, είπα και Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα ήταν ακριβώς να ε, προωθήσουν δέσμες απλούστευσης μέσω της Λισαβόνας. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι ήταν δυνατόν να αντιθέσει προς παλιές ε, προγραμματικές περιόδους να αντιδράσουμε στις ανάγκες. Και να αποφασίσουμε την τρίτη δέσμη, πράγμα που θα δώσει συγκεκριμένες ενισχύσεις για κάποια κράτη-μέλη, θα πρέπει αυτό να είναι χαρακτηριστικό και για αυτή την ε, προγραμματική περίοδο. Γιατί βέβαια και οι χρήστες χρειάζονται κάποια σταθερότητα να ξέρουν ε, ότι υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις που δεν αλλάζουν συνεχώς. Γιατί δεν είναι εύκολο να αλλάζουν συνεχώς αυτές οι πτυχές. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και με τα κράτη-μέλη πώς τροποποιείται αυτή η διαδικασία και σε σχέση με την μελλοντική περίοδο. Το ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να υπολογιστούν το προσωπικό κόστος για μικρά σχέδια νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόταν να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και σας είπα ότι στο τέλος θα έχουμε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Πρέπει συνεχώς να τη συνεχίσουμε. Αλλά έχουν γίνει πολλά νομίζω τον τελευταίο καιρό. Ναι, είμαι αρκετά ικανοποιημένο με τα όσα είπατε, Επίτροπε, και είναι άλλη μια απόδειξη για την ε, δυνητική μας δέσμευση και συνεργασία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κυρία Χιουσμένοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Χιουσμένοβα. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα είμαι σύντομη, διότι Ήδη έχετε καλύψει κάποια από τα θέματα για τα οποία θα να σα ρωτήσω. Ήδη τα έχετε απαντήσει και σας ρωτώ τώρα. Εσείς, τι θα κάνετε όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική σε σχέση με τη νέα στρατηγική της Λισαβόνα. Τι θα γίνει με την περιφερειακή πολιτική σε σχέση με τις άλλε πολιτικές της ευρωπαϊκή Ένωση, darf bei zweiterem beginnen. τη δεύτερη σας ερώτηση. Το έχω πει ήδη ορισμένες φορές. Άσχετα από τις μελλοντικές εξελίξεις, ήδη προσπάθησα να έχω κάποιες ε, συζητήσεις προσανατολισμού με δεχόμενους μελλοντικούς συναδέλφους όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους τομείς τη πολιτικής. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το προσωπικό όταν οι αρμόδιοι επίτροποι που είναι ναι, θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν δίνουμε την εντύπωση ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η συνεργασία. Υπάρχει ήδη συνεργασία μεταξύ της της περιφερειακή ε, πολιτικής και της έρευνας. Ε, συζήτησα το με τον Ιάννη Πόποτσι ε, το θέμα ότι αυτό το πνεύμα της συνεργασίας θα μπορέσει να περάσει και στον τομέα της, του περιφάλλοντος. Είχα ήδη μια πρώτη συνομιλία με τον κύριο Σιμκάρας, με την κυρία Κενβίν για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τη συνεργασία. θα πρέπει ο κάθε τομέας πολιτικής να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Άμα δούμε παραδείγματο χάρη τι επενδύουμε στον τομέα των μεταφορών πέρα από την περιφερειακή πολιτική, στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα της έρευνας, τα ποσά αυτά είναι πολύ υψηλότερα από ότι στον συγκεκριμένο εκάστοτε τομέα. Και υπάρχει το συμφέρον επίσης οι δικέ τους γνώσεις να ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική. Είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε την ολοκληρώση αυτή και όχι μια τομιακή απλώς προσέγγιση. Βλέπω ότι λείπει πάλι ο χρόνος μου, αλλά θα μπορούσαμε και αυτό να το συζητήσουμε αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Σοφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, κύριε συνάδελφοι, η περιφερειακή πολιτική πολλέ φορέ επικρίνεται διότι πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα τα οποία δίνουν οι χώρες που εισφέρουν χρήματα όπως η Γαλλία και άλλες χώρες. Σε σχέση με αυτές τις επικρίσεις δεν έχουμε μπορέσει μέχρι στιγμής να μπορέσουμε να φωτίσουμε όλα τα ωφέλη ε, τα οποία προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και έτσι να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα παντού. Εσείς μήπως μπορείτε να αναδείξετε καλύτερα αυτές τις, τις έμεσες ωφέλειες της περιφερειακής πολιτικής, δηλαδή το θετικό απότοκο αυτή τη περιφερειακή πολιτική όσον αφορά τις ε, ευρωπαϊκέ επιχείρησει από όποιον προέρχονται. Εσεί, τι πρωτοβουλίε μπορείτε να αναλάβετε ώστε να μπορέσετε να πετύχετε αυτό το στόχο. Επίση, δεν πέστε με μήπω πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ευχαριστώ. Δεν μπορούσα να απαριθμίσω όλα αυτά που πραγματοποίησε η κυρία Χίπνερ. Αλλά και αυτό είναι ένα στοιχείο. Από το 2007 ήδη υπάρχει στη Γενική Διεύθυνση ένας τομέας ο οποίος ασχολείται με την αξιολόγηση και την παρουσίαση της περιφερειακής πολιτικής. Έχετε δίκιο κυρία Βουλευτή, γιατί θα πρέπει να παρουσιάσουμε προς τους πολίτες τι πραγματοποιείται με τους πόρους που χρησιμοποιούνται εκεί. Γιατί είμαι πεπισμένος και θα το αποδείξουν και ρητά οι έρευνες, ότι και για αυτούς τους λεγόμενους καθαρούς πληρωτές η επένδυση στην περιφερική πολιτική άξιζε. Άμα δούμε τις χιλιάδες γαλλικών εταιριών που ε, έχουν άλλους ε, προϋποθέσεις σήμερα στην αγορά των μη τόσο ανεπτυγμένων ε, περιφερειών που αναπτύσσονται και έτσι οδηγούν σε θέσεις απασχόλησης στη Γαλλία. Δεν μπορεί κανένα βέβαια μέχρι το τελευταίο ευρώ να παρουσιάσει τι πληρώνει και τι εισπράττει. Παρ' όλα αυτά θα μπορούμε νομίζω να πούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από τους ε, χρησιμοποιούμενους ε, πόρους από ό,τι φαίνεται καθαρά. Καμιά φορά μάλιστα ίσως είναι επικίνδυνο να το πω αυτό. Οι λεγόμενοι καθαροί πληρωτές ωφελούνται περισσότερο από τις άλλες χώρες. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να το προσώσουμε αυτό. Είπαμε, κάν το καλό και κουβέντιασέ το κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Τεσσέρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ. Εάν εξετάσουμε το πράσινο βιβλίο για την ε, εδαφική συνοχή και για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, νομίζω πως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε χωριστά δύο ε, διαφορετικά είδη περιφερειών, τις υπερπεριφερειακές και τις μεταβατικές ε, και τις περιφέρειες μετάβασης. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα, το 75% έχουμε εκεί των κοινοτικών δαπανών θεωρείτε δυνατή τη δυνατότητα ενός προγράμματος που θα παραμένει σταθερό και θα χρηματοδοτεί τις υπερπεριφερειακές ε, περιοχές, τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, ε, για μια περίοδο μεταβατική μέσω με μιας ενδιάμεσης κατηγορίας ή για εκείνες τις περιφέρειες που πλήττονται από επίπεδο ανεργίας πολύ μεγαλύτερο από την κοινοτικό μέσο όρο. Ευχαριστώ. Also, ich habe verstanden. Εάν κατάλαβα σωστά, υπάρχει μια συζήτηση σύμφωνα με την οποία Ε, το ΑΕΠ είναι το μόνο κριτήριο με το οποίο μπορούν να γίνουν αξιολογήσεις. Γνωρίζω κάποιες συζητήσεις και η Κομισιόν είπε ότι θα συζητήσουμε κατά πόσο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι παράγοντες για την αξιολόγηση. Εγώ είμαι ανοιχτό για τις συζητήσεις αυτές. Ακόμα δεν έχουμε άλλους παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και που επιτρέπουν σε όλη την επικράτεια μια αξιολόγηση. Αλλά εάν υπάρχει πρόοδος, πιστεύω ότι η δυνατότητα θα πρέπει να τύχει τη εκμεταλλευτή μας. Όσον αφορά τις ε, περιφερειακές πολιτικές, τις, τις ε, ακραία, ακραίες περιφέρειες υπάρχουν νομίζω πολλές δυνατότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε από όσο ξέρω μέχρι στιγμής, τα μέσα που υπάρχουν είναι καλά αναπτυγμένα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον χρησιμοποιούνται επαρκώς ευέλικτα από τις περιφέρειες και από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ, Σρέντερ. Ωραία. Καλησπέρα σας, εξόδημη κυρία Χάν. Στην εισαγωγική σας ε, δήλωση είπατε, μιλήσατε για μηδενική ενοχή κατά των ε, απατών και πώς θα αντιδρούσατε αν στα μέσα ενημέρωσης υπάρχει μια κατηγορία ότι δίνονται οι πόροι αυτοί έτσι κάτω το τραπέζι θα, ε, θα δρούσατε, θα περιμένετε το ηλεκτρικό συνέδριο, θα ερχόσατε σε σύγκριση με τα κράτη-μέλη ή θα ε, δειχνόσαστε καλυμμένος όπως και στις απεργίες των φοιτητών και τι θα κάνετε αν σας κατηγορούσε το Κοινοβούλιο ότι δεν χρησιμοποιείτε σωστά τους πόρους σας. Εγώ συνήθως δεν κρύβομαι. Θα ελέγξω την κατάσταση, θα περιμένω να ασχοληθεί το ελεκτικό συνέδριο με αυτό. Πρέπει κανείς να εξετάζει κάθε κατηγορία ακόμα και αν καταρχήν ε, δίνει την εντύπωση ότι είναι αβάσιμες. Αυτό είναι κάτι που έκανα στο παρελθόν ήδη, άσχετα που είχα ευθύνη, σε ποιον τομέα δηλαδή. Αυτό είναι το στυλ μου και η γραμμή που ακολουθώ και η ευθύνη που έχω και έναντι μου του ίδιου αλλά και έναντι του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπώ. Και αυτό θα το ακολουθήσω και στο μέλλον. Δεν είναι θέμα αυτό, είναι με γι' αυτό. Είναι μια αποχρέωση εκτό αυτού που προβλέπεται από του κανονισμού μας. Συμπληρωματική ερώτηση. Στι αυστριακέ ε, ε, εφημερίδες αναφέρεται ότι υπάρχουν κατηγορίες κατά ημάν για το, τη διάρκεια της θητείας σας στην Προεδρία του Νεβαμάτικ. Κάνατε μάλιστα και κάποια δήλωση προς τον κύριο Μπαρόζο και υποβάλλατε κάθε έγγραφα, κάποια έγγραφα. Θα ήθελα να μας κάνετε και εδώ την ίδια δήλωση και να μας διαθέσετε τα ίδια έγγραφα. Ευχαριστώ, ναι, την έχω μαζί μου εδώ την... Μπορείτε να διαβάσετε μια που μιλάτε και εσείς γερμανικά όπως και εγώ. Υπήρχε απλώς μια κατηγορία ότι η εταιρεία μου αγόρασε κάποιο οικόπεδο για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν κάποια μαύρα χρήματα. Δεν έγινε αυτό. Εκτός αυτού, εγώ τότε δεν ήμουνα ούτε υπάλληλο ούτε ηγετικό τέλεχο της επιχείρησης. Μπορείτε να το δείτε και μπορείτε να δείτε ότι δεν υπάρχει καμία δικαστική έρευνα στην Αυστρία κατά του ατόμου. Ευχαριστώ. Το μας πει ο Κύριε Υποψήφια Επιτροπή, έχω δύο ερωτήσει σε σχέση με το χαρτοφυλακείο σας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρώτον, στρατηγική. Νομίζω η σχετική στρατηγική είναι δική σας και όπως νομίζετε το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα καλύψουμε μόνο εξωτερικές πολιτικές, αλλά και την περιβαλλοντική πολιτική. Για πέστε μου. Πώς θα συνεργαστείτε με όποιον αναλάβει το χαρτοφυλάκι του περιβάλλοντος για να μπορέσετε να καλύψετε και τους κινδύνους του Nord Stream για την ε, Βαλτική και το περιβάλλον της. Είχαμε ένα ψήφιμα στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2008 όπου διατυπώνονται οι λόγοι που αφορούν το περιβάλλον και θα πρέπει να σε ματέωση αυτού του έργου. Εσείς τι πρεσβεύετε σχετικά με αυτό. Δεύτερη ερώτηση για την συνεργασία σας μαζί μας. Δηλαδή την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πώς θα μας δίνετε όλο το υλικό, όλα τα έγγραφα που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία και τη χρήση των πόρων τους από τα κράτη-μέλη, τα της εκτέλεσης των προγραμμάτων και άλλων σημαντικών ζητημάτων εγώ. Ξέρετε, δυσκολεύτηκα να αποσπάσω αυτού του είδους το υλικό από από τις υπηρεσίες επιτροπής. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Για την πρώτη σας ερώτηση σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν έχω ακόμα ασχοληθεί επαρκώς. Μπορούσα να ασχοληθώ για να μπορέσω να σας δώσω εδώ μία μελετημένη απάντηση. Ξέρω το θέμα γενικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν σωστό να σας δώσω εδώ πέρα κάποια επιπόλαια απάντηση. Εάν μου χαρίσει το... την εμπιστοσύνη σας θα ασχοληθώ οπωσδήποτε αμέσω με το θέμα. Και είμαι πεπισμένος ακριβώς επειδή είδα τον Γιάννη Ποστόσικ ε, όταν ήμουν εγώ υπουργός ε, ε, επιστημών. Είναι ο συνάδελφο που ξέρω πολύ καλύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Για το δεύτερο σας ε, ερώτημα, έχετε κάθε δυνατότητα να υποβάλλετε και επερωτήσεις που θα πρέπει να αποτεθούν. Τώρα, στη λεπτομέρεια σας πω ποια έγγραφα θα σας διατεθούν και ποια θα σας διατεθούν, δεν το μπορώ, αλλά από δική μου σκοπιά έχω να σα πω ότι θέλω μέγιστο άνοιγμα. Καμιά φορά ίσως υπάρχουν κάποιες κατατάσει που για λόγους προστασίας κάποιες επιχείρησης ίσως πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικά όσον αφορά κάποιες πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά εγώ σας λέω προσωπικά είμαι υπέρ της μέγιστης διαφάνειας. Και εφόσον είναι σύμφωνο και με το, την προστασία των τομικών δικαιωμάτων θα μπορείτε να πάρετε τις πληροφορίες που σας δώσει για την εργασία σας. Thank you very much, uh, Commissioner. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ρικάρντο Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Χάν. Οι τελευταίες εκθέσεις ε, του Ελληνικού Συνεδρίου ήδη έχουν δημοσιευθεί στον κόσμο και βγαίνει μια εικόνα πάρα πολύ αρνητική όσον αφορά τη χρήση των πόρων για την ε, πολιτική που θα αναλάβετε. Το μήνυμα το οποίο παίρνει ο κόσμο, ε, δεν, δεν, έχει σχέση με την πραγματικότητα γιατί έχουμε όλες αυτές τις παραβάσεις αντικανονικότητε και τελικά δεν πρόκειται όμω για ενέργειε επιζήμιες, απλώ για κάποια λάθη. Εσεί κύριε Χάν, τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε τη διαχείριση των ταμείων αυτό να είναι όσο γίνεται πιο άρτια σε σχέση με την αρχή της αποτελεσματικότητας που πρέπει να τα διέπει. Επίση, τι άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε η ενημέρωση των, ε, των πολιτών να ε, περνάει από μια διάκριση των λαθροχειριών από τα απλά λάθη. Γιατί λάθη είναι να γίνονται λόγω του ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα σχετικά αυτά ζητήματα. Για την ερώτηση θα πρέπει ακόμα να το σκεφτώ το θέμα πολύ. Γιατί και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ που όλα σε ένα τορβανά μπαίνουν. «11» και λέγεται ότι το ποσοστό σφάλματος 11% και λεγεται οτι το ποσοστο του 11% απάτη. Αυτό ευτυχώ είναι λάθο. δεν είναι σωστό να το πούμε, παρά αυτά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, τον αντίον. Και γι' αυτό ακριβώς και η κυρία Βίμπνερ και η ομάδα της ε, υιοθέτησαν κάποια μέτρα, ούτω ώστε αυτό το ποσοστό σφάλματος να μειωθεί. Και θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια αξιολόγηση, μια έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή όπου προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου. και προσεχώς θα έχουμε την αξιολόγηση της ε, περίοδου 94-99 και θα δούμε ότι εκεί το ποσοστό πραγματικά του σφάλματος είναι κάτω από το 3%. Πολύ καλύτερο δηλαδή από ό,τι ακούμε έτσι. Το επόμενο σημείο είναι με τις αναλύσεις μας και τα μέτρα μας δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε πάντα μια καθυστέρηση κάποιων ετών. Δηλαδή γίνονται τώρα οι αναλύσεις και οι έρευνας για τα σχέδια. που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 2006 με τους όρους που ίσχυαν τότε. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα χρόνια και τα επόμενα χρόνια σε μεγαλύτερο ποσοστό θα εκλεχθούν σχέδια όπου ήδη στις προσωρινές έρευνας το ποσοστό σφάλματος είναι πολύ χαμηλότερο, κάτω από το 10% δηλαδή. Αλλά ακόμα και σας φαίνομαι εδώ αρκετά ήρεμος, είμαι πολύ ανήσυχος κατά βάση. Όπως και πολλοί από εμάς, γιατί θεωρώ ότι πολλά στην πολιτική είναι πολύ αργά. Και για εσάς σίγουρα. Αλλά οπωσδήποτε έχουν γίνει ήδη σημαντικές πρόοδοι και θα είναι και ορατή προσεχώς. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ζεμπέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Αναφερθήκατε ήδη στι ε, περιοχέ, περιοχές, αναφερθήκατε στι νησιωτικές περιοχές. Εμένα μου έλειψαν άλλε ε, περιοχέ. περιοχές. περιοχέ περιοχές και ιδίω ορεινέ περιοχές. εσεί ως ε, Αυστριακό θα ξέρετε ότι οι ορεινέ αυτές περιοχές ωραίε είναι μεν, έχουν όμως κάποια προβλήματα δε. Ε, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε κάποιο πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή νομίζετε ότι θα πρέπει οι ορεινές αυτές τις περιοχές να υπάρχουν στα αισθητικά κριτήρια όπως και οι άλλες. Ε, ως και ως Βιενέζος έχω κάποια ε, συγγένεια θέλετε με τις ορεινές περιοχές αλλά ξέρουμε και οι δύο ότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που είναι από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης. Όπως και όχι τόσο μακριά από αυτέ, υπάρχουν ορεινέ περιοχέ, οι οποίες πραγματικά είναι οι φτωχότεροι των φτωχών. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να έχουμε ευέλικτε και συγκεκριμένε αντιδράσεις ούτω ώστε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχουμε ήδη σήμερα. Πολλά ε, μπορούν να γίνουν μέσα στα πλαίσια των λειτουργικών προγραμμάτων επιτόπου. Παραδείγματο χάρη έτσι μπορούμε και σε αυτές τις περιοχές με τα ειδικά μειονεκτήματα να ε, εφαρμόσουμε τους όρους ε, των ε, περιοχών συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες και οι τοπικές δομές να προσαρμοστούν σωστά. Ich möchte da nachhaken und zwar in ερώτηση, όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε για τα κριτήρια και τους παράγοντες αυτούς, Ξέρετε ότι ιδίω καμιά φορά ε, στις ε, ορεινές περιοχές ε, οι κατακεφαλή εισοδήματα, επειδή είναι πολύ μεγάλε αυτέ τι περιοχέ, είναι πολλές φορές υψηλά. Αλλά συγκεκριμένα έχουν προβλήματα. Θα μπορέσετε να φροντίσετε τα προβλήματα αυτά να εξεταστούν συγκεκριμένα, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές είναι πολύ χοντροειδής αν θέλετε, η μέθοδος καταμέτρησης που χρησιμοποιείται. Απάντηση. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αφενό έχουμε μία συζήτηση προ την κατεύθυνση τη απλούστευση. Απ' την άλλη μεριά, προσπαθούμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για κάθε περιφέρεια κλπ. Α, καταρχήν εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε κριτήρια, παράγοντες που να είναι βάσιμα, που να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση επιτόπου. Αλλά βέβαια θα πρέπει να έχουμε 300, 300 ε, παράγοντες. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια εκτίμηση, να έχουμε κάποια εξισορρόπηση θα πρέπει η αρχή της επικουρικότητας να χρησιμοποιείται επίσης ισορροπημένα χωρίς έτσι να αυξάνομαι υπερβολικά τη γραφειοκρατία σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί θα έχουμε πανεσχέσει με τον κύριο Μπάφνερ και πόσο Ευρωπαίος είναι. Ε, Κατρίν Μπέρτερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Δεκέμβριο του 2009 η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο παρουσίασε ένα έγγραφο στην Κυρούνα, στη, Σουηδική, ε, στη Σουηδία, κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, ε, όπου ε, εξέθεται μια νέα μεθοδολογία, το MTM. Οι τοπικές αρχές θεώρησαν ότι θα ήταν μια, ένας νέος τρόπος συντονισμού και που θα ήταν ουσιώδης για την ανάπτυξη της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Αυτή η μεθοδολογία επίσης θα βοηθούσε να προσαρμοστούν οι δράσεις στις τοπικές ανάγκες και θα προσέθεταν μια πραγματικά τοπική διάσταση στις, ε, στις πολιτικές συνοχές. Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε αυτή την, ε, ε, ιδέα ώστε να αποτελέσει κεντρικό τμήμα όλων των περιφερειών αστικών και ε, γεωργικών ώστε, και πώς θα εμπλέξετε τις τοπικές κυβερνήσεις ώστε να επεξεργαστείτε καλύτερα αυτή την προσέγγιση. Απόλυτα θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή, να έχουμε δηλαδή περισσότερο περιφερειακές τοπικές δομές και να προσπαθήσουν και μέσα στα πλαίσια της εταιρική σχέσης να εμπλέξουμε και μη κυβερνικέ οργανώσεις, εκπροσώπηση της ε, κοινωνίας των πολιτών. Να έχουμε κάποιες συγκεκριμένε ε, ε, δυνατότητες γιατί η πολυμορφία της Ευρώπης ξεκινάει από την πολυμορφία των τοπικών και περιφερειακών της δομών και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Thank you. Um, in particular, my... Σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερα η δική μου περιοχή της νοτιοανατολικής Αγγλίας είναι ευημερής και ίσως να μην ε, θεωρείτε ότι χρειάζεται στήριξη. Ωστόσο, φιλοξενεί πολλούς ε, κινούμενους εργαζόμενους από την Ανατολική Ευρώπη και τα τοπικά συμβούλια και οι τοπικές αρχές προσπαθούν να στηρίξουν αυτούς τους ε, κινούμενους εργαζόμενους και θα ήθελα να δω πώς μέσω των LDM μπορείτε να στηρίξετε αυτές τις πιο ευημερείς περιοχές και πώς μπορείτε να παρεμποδίσετε τα εμπόδια που προκαλούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, ε, ορισμένοι θα το ονόμαζαν αυτό παρέμβαση των κρατικών κυβερνήσεων στις ενέργειες των τοπικών αυτών αρχών. Ναι, καλή ιδέα. Ε, διακυβέρνηση πολυεπίπεδη θα λέγαμε αλλά καταρχήν θα πρέπει εμείς ως Επιτροπή να αναζητήσουμε τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αλλά στον διάλογο αυτό με τα κράτη-μέλη, όσον αφορά τις στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές κλπ, θα πρέπει και θα φροντίσουμε, και το κάναμε ήδη στο παρελθόν, να έχουμε κατά νου ενδυναμωμένη τοπική ένταξη Εσείς αναφερόσατε εδώ κυρίως ε, στο Διευθυντικό Ταμείο που είναι κάπου εδρεωμένο ε, σε εθνικό επίπεδο και ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουν να χρησιμοποιούνται οι πόροι πιο περιφερειακά, πιο συγκεκριμένα, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση από τις ε, τοπικές, από τις περιφερειακές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βίκτορ Μπουστινάρ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφιο επίτροπε. στι απαντήσει προ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρατε μεταξύ των πιο σημαντικών πρωτοβουλειών που θα αναλάβετε κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων ω επιτρόπων την ε, στρατηγική για το Δούναβι. Εμεί, στην Επιτροπή Ρέτζι και εγώ ίδιο ω ρουμάνο, ε, καλωσορίζω ιδιαίτερα αυτή την δέσμευσή σα και την πρωτοβουλία σα για, πρωτο... για πρόθεση αυτή τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικέ σας, ε, οι στο σχεδιασμό σχεδιασμό της στρατηγικής, όπου φυσικά το Κοινοβούλιο θα είναι εταίρος σας και φίλο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς, αυτή η τελευταία παρατήρηση ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο αυτό. Γιατί αφορά αφορά κράτη-μέλη και έξι χώρες που δεν είναι ακόμα ε, κράτη-μέλη. Και από δική μου σκοπιά, πρόκειται για ένα πολύ θετικό μήνυμα σε σχέση με μια μακροεδαφική συνεργασία όπου ο Δούναβης είναι ο συνδετικός κρίκος αν θέλετε. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουν πρώτα σεμινάρια όπου μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να καθοριστούν τα κεντρικά σημεία και ελπίζω πολύ από εσά να συμμετάσχετε στις δραστηριότητε αυτές, να συμβάλλετε και έτσι στα πλαίσια του προγραμματισμού του σχεδίου να ε, συμβάλλετε σε αυτή τη στρατηγική για το Δούναβι. Μου φαίνεται ο σε σχέση με την πολιτική ΟΣΕΑΜ είναι η δεύτερη σημαντική προσπάθεια σε συνεργασία με περιφέρειες που έχουν παρόμοια προβλήματα παραδείγματο χάρη για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση πλωτών οδών να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα συνεργασία, παραμένοντα βέβαια στι αρχικέ ιδέες ότι θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικέ δομέ δεν θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάντα βασιζόμενοι στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει για τις εν λόγω περιοχές. Thank you very much Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πεπισμένοι ότι εάν την επομένη εβδομάδα περάσει αυτό το ψήφισμα όσον αφορά την μέλου στρατηγική της ΕΕ για τις νέες περιφέρειες, πρόκειται να έχουμε μια πολύ σωστή αφετηρία. Εσείς ως Επίτροπος και εμείς ως Κοινοβούλιο, οπότε έτσι θα έχουμε δεσμευτεί για μια συνεργασία παραγωγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιώσιφ Ματούλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια, Επίτροπε. Στην προηγούμενη απάντηση μας αναφέρατε ότι η πολιτική της συνοχής ε, αποτελεί ακόμα ένα επίπεδο σύγχρονο, ε, μοναδικό επίπεδο διακυβέρνησης, το οποίο βασίζεται ε, στη γνώση των τοπικών αρχών και ότι βοηθάει όσον αφορά τον συντονισμό των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνηση. και είπατε ότι στο μέλλον θα ενδυναμωθεί αυτή η κατάσταση, θα ενισχυθεί και επίση ε, θα αναδειχθεί το πόσο σημαντική είναι η τοπική παράγοντε. Και κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται να έχουμε και ίσως και άλλες παραλλαγές ε, τοπικής περιφερειακής οργάνωσης ή στο μέλλον σε σχέση με την πολιτική συνοχή, πώ όλα αυτά θα, θα, θα εμπλέκονται, ε, ποιο, ποιο όργανο, ποιο επίπεδο θα έχετε τον πιο σημαντικό ρόλο. Η προσέγγιση βέβαια κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορεί να είναι. Μην το έχετε σκεφτεί αυτό. ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη θα υπάρχει ενιαία διοικητική δομή. Γιατί όπως είπαμε, ακριβώς η πολυμορφία, η, χάρη της Ευρώπης είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις που οδηγούν σε διαφορετικές ε, κρατικές μορφές οργάνωσης. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια των δομών αυτών στην Ευρώπη. Πώς θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη ευελιξία. Πώς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιο είναι εκάστοτε το κατάλληλο όργανο με το οποίο θα μπορέσω να ζητήσω τη συνεργασία. Χρειάζεται λοιπόν ε, ευέλικτη δράση και αντίδραση, αλλά θα πρέπει μέσα στα πλαίσια των ε, επισήμων δομών να είμαστε ευέλικτοι επαρκώς, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και άλλες δομές. Η περιφερική πολιτική μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν εμπλακούν οι πολίτες. Δεν υπάρχει καμία πολιτική στην οποία οποία η Ευρώπη είναι τόσο ορατή, τόσο κινδυνεύει θα έλεγα κιόλα όμως και είναι ευάλωτη όσο η περιφερειακή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι πρέπει. Καλούνται οι υπεύθυνοι να δείξουν κατά το δυνατόν μεγάλη ευελιξία και για την συνεργασία των πολιτών και να μην ε, αναφερθούν υπερβολικά σε ε, τυπικές δομές. Μαρία Τερέζα transfrontalière un de premier plan Αυτή η πολιτική σα ωφελεί εκατομμύρια Ευρωπαίων. Αφορά και τι όμορε χώρε, Πρόκειται μια πολιτική η οποία έχει άμεσα αποτελέσματα. Πρόκειται για κάτι το οποίο για σας είπατε ότι έχει προτεραιότητα, αλλά στην πολιτική συνοχής πώς εντάσσονται όλα αυτά, τι θα κάνετε σε, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα για την πολιτική αυτή. Κοιτάξτε, μάθαμε από την ιστορία μας και πρέπει να το μάθουμε ότι το χειρότερο είναι να ε, σκεφτόμαστε σε σύνορα και να ε, κινούμεθα σε σύνορα. Δεν το κάναμε ευτυχώ και γι' αυτό είμαστε τόσο ισχυροί και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε κάθε πολιτική που ξεπερνάει τα σύνορα. Ό,τι και αν εννοούμε υπό την έννοια σύνορα. Κατά πόσο να πρόκειται σύνορα μέσα σε μια περιφέρεια, μέσα σε μια χώρα η περιφερειακή συνεργασία περισσότερων περιφερειών, κατά πόσον έχουμε μια συνεργασία μεταξύ μεθοριακών περιοχών στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν πρόκειται για συνεργασία ευρωπαϊκών περιφερειών με περιφέρειες συνοριακών ε, τρίτων χωρών. Θα πρέπει πάντα να προωθήσουμε τη συνεργασία αυτή, να την υποστηρίξουμε, γιατί αυτό είναι μια πολιτική την οποία εγώ προασπίζω, μια που πιστεύω ότι είναι η μόνη δυνατή πολιτική για να πετύχουμε μια προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ευμάρια, κράτος δικαίου και πολιτική σταθερότητα σε άλλους τομείς εκτός της Ευρώπης. Vous dites que les frontières ne doivent pas être des obstacles, mais euh, pensez-vous que l'échelon européen peut agir pour... Κοιτάξτε, πιστεύετε πως ε, θα μπορείτε να λάβετε μέτρα για να αντιμετωπίσετε τη στρέβλωση της αντικονιστικότητας που υπάρχει στις όμορες ε, χώρες, ε, καθώς επίσης και ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Ειλικρινά, αυτή είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εάν δεν το πίστευα αυτό, αν δεν είμαι πεπισμένο γι' αυτό, ε, τότε δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Είμαι πεπισμένο 100% ότι αυτού του τύπου η πολιτική μπορεί κάτι να αλλάξει. Μα ακριβώς εγώ ασχολούμαι με την πολιτική επειδή ήθελα κάτι να καταφέρω, κάτι να αλλάξω. Και η διαμεθορική συνεργασία Ιδίω, αν σα κατάλαβα σωστά, με τις περιφέρειες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οπωσδήποτε κάτι που θα πρέπει να προωθήσουμε. Και στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της Ιδρυτικής συνθήκης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη κυρίως είναι ένα σχέδιο ειρήνης και θα πρέπει αυτό να το προωθήσουμε και περαιτέρω και θα πρέπει να το ασπαστούμε επίσης. Και άμα υπάρχουν κάποια διακυβερνικά προβλήματα ή προβλήματα ε, διοίκηση θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, στο πλαίσιο των νέων παγκοσμίων προκλήσεων που είναι και ε, κοινοτική και περιφερειακή και προκλήσεις ή ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές πέρα από τους ε, ιδιαίτερους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται έχουν τεράστιες δυνατότητες που κυρίως στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων μπορεί να δώσουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για αυτές τις ε, περιφέρειες που όχι μόνο βέβαια διατηρούν την ε, τις δυνατότητές τους, αλλά μπορούν να βάλουν στην υπηρεσία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ε, δυνατότητες αυτές που έχουν. Absolut, Sie laufen bei mir hier offene Türen ein. Ähm, εγώ μπορώ απλά να επαναλάβω αυτό που είπα μόλις τώρα. Δεν εννοώ την πολιτική εγώ ως την δυνατότητα να επιβάλλω σε άλλους το δικό μου τρόπο ζωής. Και να πω, όπως εγώ ζω πρέπει να ζουν και όλοι οι άλλοι. Όχι, τον αντίον. Απ' την άλλη μεριά μας αυτό για το οποίο είμαι σε 100% είναι ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο ζωής είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Είναι ένα πρότυπο για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι και που ε, κάπως μπορούμε να το παρουσιάσουμε και σε άλλους. Το τι θα κάνουν οι άλλοι τώρα με αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν οι ίδιοι. Εγώ δεν μπορώ να τους ε, πιάσω το λαιμό και να τους πω ότι θα κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς. Όχι. Αλλά θέλω πολύ να γνωρίσουν καλύτερα το δικό μας μοντέλο, να ξέρουν τι μπορέσαμε να κάνουμε και ιστορικά και τι μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον. Πολλά μπορεί να καταφέρει το ευρωπαϊκό μοντέλο και γι' αυτό πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες σαν αυτή που περιγράψατε θα πρέπει να τις συνεχίσουμε. Πρέπει να έχουμε την υποχρέωση έναντι ημών αλλά και άλλων όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε για την εργασία, για την ζωή. Όλα αυτά να τα κοινοποιήσουμε και σε άλλους ελπίζοντας ότι θα το ε, επομισθούν. Αλλά η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από εκείνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σαν Κέλλη. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, η πολιτική συνοχή και η πολιτική μεταφορών συνδέονται στενά μεταξύ τους και προγράμματα όπως το τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική συνοχή. Μιλήσατε, για την οικοδοκατασκευή εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων που μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Ως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, πώς προβλέπετε την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς ε, δράσεις, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την βιώσιμη πολυτροπική, τις, μάλλον, τις υποδομές για την βιώσιμη πολυτροπικές μεταφορές ε, και όλα αυτά με ιδιαίτερη αναφορά στις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και την άλλη της διαστάσεις ε, της περιφερειακής ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι πολύ προσφυλή σε εσάς, αν κρίνουμε από τις αρχικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Yeah. Genau Ακριβώς ε, πάνω στο θέμα αυτό είχα μια πρώτη συζήτηση ε, μετά από πρόσκληση του Συμπάλα, ε, Κάλλας μάλιστα, για το θέμα ότι πώς μπορούμε οι, οι υποδομές μεταφορών στον αστικό τομέα να βελτιωθούν από κοινού. Γιατί νομίζω όλοι μας έχουμε ντουζίνες, να μην πω εκατοντάδες παραδείγματα. Ακόμα και στον περιφερικό τομέα. Δηλαδή μεταφορές μεταξύ της πόλης στο κέντρο και της ε, ε περιφέρειάς της. Ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ε, δυνατότητα μεταφοράς ε, Πρέπει να υπάρχει συντονισμό. Εγώ δεν αφαίνομαι εδώ πέρα στα διευρωπαϊκά δίκτυα, όπου πάλι καλούμεθα ως ε, ε, περιφερειακή πολιτική να δράσουμε στην Την model split. Νομίζω ότι ακριβώς στις αστικές περιοχές χρειάζεται να δράσουμε και πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν και υπό τη σκοπιά της βελτίωσης της χρήσης ενέργειας, των κλιματολογικών αλλαγών. Αν καταφέρουμε οι αστικές μεταφορές να είναι ιδανικότερες και έτσι να συμβάλλουμε ούτω ώστε παραδείγματο χάρη όσον αφορά τους εργαζόμενους να γίνεται καλύτερη, ακόμα καλύτερη εκμετάλλευση των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Αλλά εδώ θα πρέπει να υπάρχει βέβαια και η διαθεσιμότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής. Και θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας να μην σπαταλάτε κατά οποιοδήποτε τρόπο η ενέργεια ακριβώς στα αστικά κέντρα. Είμαι ευχαριστημένος στην απάντησή σας και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να θέσω σε αντίθεση με τους κανόνες ε, δεν θα κάνω λοιπόν επερώτηση. Ο κύριος Χαράλαμπος Αγκουράκης. Πού βρίσκεστε? Uh, Δεν... είναι εδώ ο συναδελφός μας. Οπότε περνάμε στον Τζον Μπάφτον. Σα um, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι. Κύριε Χάν, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο πρόσφατα δήλωσε ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι υπεύθυνε για το μεγαλύτερο ε, κομμάτι των ε, σφαλμάτων ε, όσον αφορά τα περιφερειακά, την περιφερειακή ενίσχυση. 2,7 δις ευρώ λείπουν. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε τι μέτρα θα χρησιμοποιήσετε κατά αυτών των τριών χωρών. Ειλικρινά, θα εξετάσω τις λεπτομέρειες του θέματος. Εγώ δεν μπορώ και δεν θα ήθελα σήμερα να βιαστώ με κάποια δήλωση, γιατί ακριβώς δεν έχω τα ακριβή στοιχεία στα χέρια μου. Ξέρω ότι από πλευράς της Γενικής Διεύθυνης Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν λάβει χώρες συγκεκριμένε διαβουλεύσεις με τις εν χώρες και θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αυτών που είναι σφάλματα ή εκείνων που λαμβάνουν χώρα μέσα στα πλαίσια κάποιων ε, δημοσιονομικών διορθώσεων. Και ακριβώς τα τελευταία χρόνια υπήρχε σημαντική ανάπτυξη των διορθώσεων αυτών. Το 2008 και 2009, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2,5 δις ευρώ το ύψος των διορθώσεων αυτών. Πολύ σημαντικό ποσό πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνουν υπόψη μας αυτό το μέτρο. Αλλά ξαναλέω, ο στόχος μιας περιφερικής πολιτικής δεν είναι στο τέλος της ε, προγραμματικής περίοδου να μπορώ να πω εξοικονομήσαμε χι δισεκατομμύρια, δεν τα δαπανίσαμε καθόλου. Ο κοινό μα στόχος θα πρέπει να είναι τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται στις περιοχέ σύμφωνα με τι συμφωνίε που έχουν υπάρξει για τα εν λόγω προγράμματα. Δεν μπορεί ο στόχος μας της περιφερειακής πολιτικής να είναι να πούμε τελευταία αναλήξη. Θαυμάσια, ξεκονομήσαμε χι χρήματα. Τι ωραία που δεν τα ταπανίσαμε. Όχι, όχι. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των πολιτών και να χρησιμοποιηθούν σωστά και προς όφελος των πολιτών που είναι φορολογούμενοι. Και από ό,τι βλέπουμε από τα στοιχεία βλέπουμε ότι υπήρχαν σημαντικές βελτιώσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Well, Uh, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστια τα ποσά. 2,8 δις ευρώ δεν είναι και μια σταγόνα στον ωκεανό, είναι ένα τεράστιο ποσό. Και ελπίζω να συμφωνείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, να μπορώ να σας αποκαλέσω ακόμα έτσι για τον προπολογισμό και τις ιδέες σας για τον προπολογισμό. Όπως ξέρετε υπάρχει μια πρόταση προπολογισμού που προβλέπει ε, ουσιαστικό περιορισμό του Ευρωπαϊκού Δομίου Περιφερειακής Ανάπτυξης μεταξύ των άλλων και διαγραφή των στόχων στόχου 2, των σχεδίων συγγνώμη στόχου 2. Η ερώτησή μου ποια είναι η στάση σε αυτό και στο μέλλον θα μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι στο μέλλον θα ωφελούνται από το Ταμείο Συνεχής και φτωχότερες ε, περιοχές λεγόμενων καθαρών πληρωμών. Ναι. Για την τελευταία ερώτηση έχω να πω ναι. Καταρχήν επαναλαμβάνω. Η περιφερική πολιτική είναι προς όφελος όλων των περιφερειών της Ευρώπης. Αυτό που αναφέρατε ήταν κάποιες σκέψεις που άρχισαν να κυκλοφορούν γραπτά. Θα πρέπει να χαιρόμαστε που υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, γιατί μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν μόνο εκείνοι που είναι υπέρ της πολιτικής μας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κριτική. Σωστό μου φαίνεται. Και σας λέω επίσης ότι εγώ είμαι υπέρ μιας πολιτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης περιφερειακής πολιτικής. Όχι μόνο για να κάνω εντύπωση επειδή είμαι ε, υποψήφιος τώρα ως ε, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, αλλά το είχα κάνει και στο παρελθόν και τώρα μάλιστα μελετώντας το υλικό εις βάθος είμαι πεπισμένος ότι μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Επαναλαμβάνω, πάντα όμως συμπεριλαμβάνοντας και όλους τους άλλους το της πολιτικής. Θα ήταν πάρα πολύ ασφαλμένη η προσέγγιση να θεωρούσαμε ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι, ό,τι θέλει και ότι η περιφερειακή πολιτική είναι ε, μια μορφή τομιακής πολιτικής. Θα ήταν μοιραίο να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, καταστροφικό. Και από μέχρι τώρα συζητήσεις με τους ενδεχόμενα μελλοντικού μας ε, συναδέλφους, βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτού του είδους το σκεπτικό. Ότι ο καθένας ασχολείται δηλαδή με το δικό του τομέα. Αλλά ότι υπάρχει κατανόηση ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση 2020 και εκεί θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε και η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Τελευταία παρατήρηση. Ακριβώς αυτή τη στιγμή που για πρώτη φορά η περιφερειακή πολιτική έχει εδρεωθεί στη συνθήκη μέσα στα πλαίσια της ε, περιφερειακής ε, συνοχής. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουμε την ιδέα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι κάπως διαφορετική. Κύριε Υπουργέ, από το 1997 ως το 2003 ήσασταν πρόεδρος ε, μιας επιχειρήσης Novomatic και σε κάποιον από του ε, συναδέλφου είπατε ότι δεν υπάρχει καμία ε, προσφυγή κατά τις εταιρείε αυτές. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια προσφυγή λόγω φοροδιαφυγής. Ίσως δεν υπάρχει πια, θα το χαιρέτιζα. Αλλά μήπως αυτό ίσως επιβαρύνει την εργασία σας ως επιτρόπου. Μισό λεπτό. Δεν είναι υπερώτηση. Οπότε ε, ο Επίτροπος μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Αλλά είναι πάντως ε, ε, ενάντια στους κανόνες μας. Απλώς θέλω να σας το πω αυτό. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Εγώ είπα κατά εμού δεν υπάρχει καμία προσφυγή. Αλλιώς δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά για μένα. Κατά εμού δεν υπάρχει καμία έρευνα δικαστική ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, Καρή Μαντελή. Στα αριστερά κάθετε. Καλησπέρα σα, κύριε Αν. Αν δούμε του στόχου τη στρατηγική τη Λισαβόνα, δηλαδή να γίνει πιο ανταγωνιστική οικονομία, περισσότερη απασχόληση, περισσότερη κοινωνική συνοχή και το βασικό στόχο τη μείωση τη φτώχεια το 2010, ενώ φτάνουμε στο τέλο, ε, είμαστε πολύ μακριά όσον αφορά ε, τον αγώνα κατά τις στόχες. Δεν την έχουμε κερδίσει την μάχη αυτή. Στο Βέργιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία υπάρχει μέγας κίνδυνος γι' αυτό και για τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και κυρίως για τους νέους. Οι πολιτικές συνοχές θα μπορέσουν να αντιστρέψουν αυτή την τάση και να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις, γνωρίζοντας ότι το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις πόλεις που θα δεσμευτείτε για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή στο πλαίσιο των αστικών ζωνών Δαπανών αποτελεί προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ja, das muss eine Priorität darstellen. Ε, πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Ιδίω ε, εδώ είναι σημαντική συνεργασία με την συναδελφό άνθρωπα. Θα πρέπει να αντιστοιχθεί εκ μέρου μου. Θα το κάνω αυτό και ξέρω ότι μέσα στα πλαίσια του Διευθυντικού Ταμείου, ιδίω ε, λόγω της οικονομικής κρίσης, υιοθετήθηκαν γλίγορα και ευέλικτα μέτρα, όπου κατεβλήθη ακριβώς προσπάθεια αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. και είδα ας πούμε ότι σε πολλά κράτη ε, υιοθετήθηκαν κάποια μέτρα, διαθέθηκαν συμπληρωματικοί πόρη, κατεβλήθη προσπάθεια γρήγορης αντίδρασης. Ε, το άμεσο έργο του Ζωδιαθωτικού Ταμείου δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δράσει για την γενική ανάπτυξη. Ε, βέβαια, ειδικέ καταστάσεις απαιτούν ειδικά μέτρα. Euh, une question supplémentaire. Euh. Ε, επέρωτης. Το πρωί ο κύριος Σέτιγκερ, ο μέλλον της άνθρωπος, είπε ότι θα δοθούν περισσότερα χρήματα τόσο ώστε να υπάρχει βελτίωση ενεργειακά των κτηρίων. Χρήματα από τα διαφορετικά ταμεία. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση αυτή του συναδέλφου σας. Ούτως ώστε με διαρκή τρόπο να σταματήσουμε να έχουμε ενεργειακή ανασφάλεια για όλη την Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι δυνατό λόγω της δέσμη απλούστευσης, όπως λέμε. Τώρα θα δούμε, θα εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητε ή όχι. Ελπίζω ότι θα τύχει εκμεταλλευση σε μεγάλο ποσοστό. Uh, uh, Κύριε Χάν, φορείς, τοπική, περιφερειακή, δήμοι, κοινότητες ζητούν πιο αποφασιστική στάση όσον αφορά την πολιτική της συνοχής. Εσείς, τι λέτε, κάτι τέτοιο είναι θετικό για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Στέκει το να μιλούμε για αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. εάν οι πόλεις και μικρότερες ε, μονάδες ε, συμβάλλουν στην ε, πολιτική συνοχή. Σε αυτό ήταν το ερώτημά σας. Ζητούν πιο αποφασιστικές τοποθετήσεις, θέσεις, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εποπτεία, την δηλήψη των αποφάσεων, την αξιολόγηση. Και σας ερωτώ, Είναι θετικό ή αρνητικό αυτό που ζητάνε κάτι εσά. Θετικό μου φαίνεται. Γιατί και εδώ έχουμε αυτή την ε, σκέψη της ε, επικουρικότητας. Εάν το λάβουμε σοβαρά υπόψη, το θέμα της επικουρικότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί κιόλα. Ίσως καμιά φορά στην πρακτική εργασία ε, είναι κάπως κουραστικό γιατί πρέπει να υπάρχει συνονισμός με πολλούς. Από την άλλη μεριά είμαι πεπισμένος και λόγω της μέχρι τούδε πολιτικής μου δραστηριότητας ότι καμιά φορά διαρκεί περισσότερο το να καταλήξουμε σε αποφάσεις και εκτιμήσεις, αλλά όσο πιο πολύ συμμετά έχουμε εδώ, τόσο πιο αηφόρες είναι οι αποφάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς όπως ήταν και η συζήτηση με τους καθαρούς ε, πληρωτές. Κάτι δηλαδή όπου υπάρχει αυξημένη ε, προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα δικαιολογεί τις συμπληρωματικές αυτές προσπάθειες. Το ξέρουμε όλοι αυτοί ότι όταν επιβάλλουμε την άποψή μας σε κάποιους, βραχυπρόθεσμα ίσως είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι εις βάρος αυτών που επέμειναν έτσι. Γι' αυτό λέω ναι, σε πιο έντονη συνεργασία γνωρίζοντας ότι αυτό δεν διευκολύνει την εργασία, αλλά γνωρίζοντας επίσης ότι εν τελευταία αναλύση θα ωφεληθούμε όλοι. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Σήμερα τηρήσατε πολύ αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές και του Προέδρου Μπαρόζο εδώ και πολλά χρόνια ήσασταν και μέλος της ε, αστικής κυβέρνησης ε, της Βιέννης. Είσαστε δηλαδή σε μια μητρόπολη υπεύθυνο και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω ε, θα έπρεπε να, να αναφερθείτε περισσότερο στην ανάγκη της πρόθεσης της ε, τοπικής και επίσης αναφερθείτε στην καινοτομία χωρίς να μας πείτε τίποτα συγκεκριμένο. Θα ακολουθήσετε μια καινοτομική πολιτική όσον αφορά παραδείγματος κάνει την ίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι καλό θέμα αυτό στην Ευρώπη. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι εδώ, γιατί έχουμε περισσότερες χώρες μέλη, έχουμε περιορισμένους πόρους, λιγότερους πόρους ίσως από ό,τι παλαιότερα. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε καλύτερα λοιπόν αυτό που εννοείτε. Αναφερθήκατε ε, στο περιεχόμενο ε, αφενός και ε, στην άλλη κατά πόσον θα πρέπει περισσότερο να χρησιμοποιηθούν νέα χρηματοδοτικά μέσα. Και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποιες πρώτες πρωτοβουλίες. Εγώ τις χαιρετίζω αυτές ρητά. Κατανοώ επίσης ότι στο επίπεδο των τομέων αυτών της ε, μελλοντικής πολιτικής θα έχουμε την εμπιστοσύνη να ασχοληθούμε με το θέμα. Γιατί είμαι πεπισμένος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς ότι σαν καινοτομική προσέγγιση με πεπισμένος λέω ότι θα πρέπει από μία πολιτική δωρεών να περάσουμε σε μία πολιτική δανείων, διότι έτσι θα υπάρχει και πιο έντονη δέσμευση των δικαιούχων για κάποια συγκεκριμένα σχέδια και έτσι θα υπάρχει και δυνατότητα επίδρασης πολύ εντονότερη με τους πόρους αυτούς να πραγματοποιήσουμε πολύ περισσότερα σχέδια. Μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια πολύ καινοτομική προσέγγιση αυτή. Αν μπορέσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επίσης, να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, μικροδάνεια παραδείγματο χάρη, και εδώ υπάρχουν κάποιες πρώτες ε, πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Αλλά θα μπορούσαμε έτσι να αναπτύξουμε τα σχετικά μέσα γιατί καμιά φορά στη, οι τίτλοι είναι πολύ ωραίοι, αλλά στην ε, εφαρμογή βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Αλλά εδώ θα θέλω να κινηθώ, γιατί νομίζω ότι ο χρόνος έχει πραγματικά φτάσει να το κάνουμε και εκτός αυτού το χρειαζόμαστε απαραίτητα. Ευχαριστώ. Μια συμπληρωματική ερώτηση. Ακριβώ αυτή την κατεύθυνση θεωρούσα και εγώ ότι δεν μπορούμε κανένα, να, να ραντίζουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί, σε όλου του τομεί Ευρώπη. Και άμα κοιτάξουμε το 98% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Ε, και θα ήθελα να ρωτήσω, προτίθεστε πραγματικά να ενισχύσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με περιφερειακά σχέδια. Τεχνολογία, παραδείγματος χάρη, είναι η πρόθεση διάφορων κλάστερς. Ε, προτίθεστε να κινηθείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Στα πλαίσια του θέματος έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, ναι. Αυτό είναι που λέω. Υπάρχουν μεγάλες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει κανένας πραγματικά να κινηθεί. Και αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, έχω κατά νου παραδείγματος ένα αριθμητικό στοιχείο που λέει ότι στην περασμένη προγραμματική περίοδο μόνο για τη Γαλλία υπήρχαν 13.000 επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν στον τομέα της καινοτομίας. Κάτι έγινε λοιπόν. Κάτι γίνεται λοιπόν. Από τους πόρους που έχουμε ήδη δίνουμε 86 δισεκατομμύρια ευρώ για όλο τον τομέα της καινοτομίας όπου σήμερα ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ήδη δηλαδή πολλά γίνονται και αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί στο μέλλον. Βέβαια πάντα αναβάνουν υπόψη τις μεγάλες στρατηγικές κατευθύνσεις γραμμές. Και στην Βεστιβάλα. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αστική διάθεση, στην, διάσταση στην περιφερική πολιτική, κύριε Χάν θα ήθελα να πω ότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μένες ζουν στο αισθητικό επίπεδο. Ε, θα ήθελα να δούμε ότι υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Αναφερθήκατε σε αυτά, δημοκρατική αλληλεγγύη. Εκτός αυτού, οι πόλεις έχουν βέβαια ένα ιδιαίτερο ρόλο να παίξουν όταν πρόκειται να βελτιώσουν του όρους διαβίωσης των πολιτών. Και εδώ υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια από μέρους όσον αφορά την ανάπτυξη των πόλεων μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής, συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή, οι σχέδια και πώς μπορούν οι πόλεις αυτές συγκεκριμένα να συμπεριληφθούν στην ε, αστική εξέλιξη και μπορείτε να φανταστείτε ότι οι περιφέρειες θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία αναφέρατε. Θα πρέπει να σας πω ότι και για τις ε, πόλεις, όπως και για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρώπης, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως υπάρχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ε, το αυτό και με την εμπειρία την οποία έχω, δεν θα ήθελα να πω τι μπορούμε να κάνουμε στις πόλεις, γιατί έχω την εμπειρία της Βιέννης και η κατάσταση σίγουρα είναι παρόμοια ε, και σε άλλες πόλεις. Άλλες πόλεις της Ευρώπης, λό με βέβαια με διαφορετικούς όρους ε, και λόγω διαφορετικών ιστορικών εξελίσσεων, έχουν και κάπως... Ε, αντιμετωπίζουν και κάπως διαφορετικά προβλήματα. Στη Βιέννη, για παράδειγμα, ε, ε, εμείς ε, μιλήσαμε για τη χρήση των επιφανειών στο κέντρο της πόλης, προβλέποντας να καλύψουμε τον σταθμό για να έχουμε παραπάνω χώρο. Σε άλλες πόλεις ε, το πρόβλημα είναι ας πούμε ο ανεφοδιασμός σε πόσιμο νερό. Ήδη έχουμε μιλήσει για το πρόβλημα των μεταφορών. Πάντως αυτό που είναι προφανές και αυτό που το γνωρίζουμε είναι το, ότι το 80% των Ευρωπαίων ζουν ε, σε αστικές περιοχές. Ε, δεν θα έλεγα πως όλες αυτές οι αστικές περιοχές είναι πόλεις και θα πρέπει σίγουρα και οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με αυτές. Δεν θα είναι δυνατόν να υποχρεώσουμε τις περιφέρειες σε κάτι Μιλήσαμε ήδη και επανέρχομαι σε αυτό ότι δηλαδή Εάν συγκεντρώσουμε έναν μεγάλο αριθμό συνομιλητών μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα που ξεπερνούν τις ε, τυπικές αρμοδιότητες στην περιφέρεια της Ανατολικής Αυστρίας για παράδειγμα και το αναφέρω αυτό ε, ως ε, παράδειγμα καταφέραμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο μεταφερών δεν μπορέσαμε δικτύως δυστυχώς να φτιάξουμε και άλλα δίκτυα αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλες τις πόλεις ε, μαζί με τις περιφέρειες που τις ε, περικλείουν και ίσως και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο των συζητήσεών μας στους επόμενους επόμενους ε, Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να προωθήσουμε την επιθετική πολιτική των πόλεων ε, ε, οδηγώντας και τις περιφέρειες σε συμμετοχή σε αυτές τις πολιτικές. Πιστεύω πως αυτό που οι πόλεις επιθυμούν να ακούσουν είναι ότι ως πολιτικοί θέλουν πραγματικά να ενταχθούν και να εμπλακούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μωρίς Πόγκα, πού βρίσκεσαι? Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές που είναι, όπως το είπατε, στις αρχικές σας δηλώσεις που εμπλουτίζουν την Ευρώπη. Γνωρίζετε τι νέε προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες όπως η παγκοσμιοποίηση και οι κλιματικέ αλλαγέ, και οι περιφέρειες μα αποτελούν ε, τι πιο ευάλωτε περιφέρειες απέναντι σε αυτές τις νέε προκλήσεις. Μπορείτε σε αυτό το πλαίσιο να μα δώσετε τη θέση σα όσον αφορά την κατανομή των αντισταθμίσεων του παραπάνω κόστου που συνδέεται με τον ισχυρικό χαρακτήρα και την απομακρυσμένη του γεωγραφική θέση ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε με περισσότερο περισσότερη ψυχραιμία τους μεγάλους προσανατολισμούς των περιφερειακών ε, πολιτικών και να εκμεταλλευτούμε τα τούτους που ήδη είναι ε, αναγνωρισμένα. Also, ich würde sagen, dass äh, schon bisher äh, von Seiten der Europäischen Union ε, Ήδη σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και δημοσιονομική στις ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιοχές. Και αυτή η προσοχή αντοκατοπτρίζεται και στην ε, συνθήκη. Πιστεύω λοιπόν πως ε, έχουν τεθεί στους κατάλληλες βάσεις για το μέλλον. Αντίθετα και δεν αποφεύγω το ερώτημά σας, όλα τα θέματα που συνδέονται με τα οικονομικά, δεν μπορούν απαραίτητα να χρηματοδοτηθούν από την περιφερειακή πολιτική. Υπάρχουν ε, πολιτικές ε, ενίσχυσης με διαφορετική διάσταση. Ωστόσο, εγώ είμαι υπεύθυνο για τις ε, πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές και άρα την κατάλληλη στιγμή, όταν αυτό χρειαστεί, θα παρέμβω. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην περιφερειακή πολιτική και την ε, βοήθεια προς τις περιφέρειες και της ε, γενικότερης πολιτικής ενισχύσεων με άλλους στόχους. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάντενμπαχ, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα άμεσα να επανέλθω στην τελευταία σας παρατήρηση. Στην αρχή της ε, σημερινής σας ε, δήλωσης είπατε ότι είστε ο πατέρας των περιφερειών. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι είμαι μητέρα ε, πέντε παιδιών και πιστεύω ότι θα πρέπει να παρεμβαίνει κανείς εκεί όπου πρέπει να εξαλείψει τα ελλείμματα και να ενθαρρύνει αντίθετα τα ταλέντα σε όλα τα ερωτήματα που θέσατε συμφωνήσατε μαζί μας, αλλά γνωρίζουμε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς το σημερινό προπολογισμό και τις σημερινές πιστώσεις. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τις αυξήσουμε και ότι οι πιθανότητες να τις αυξήσουμε είναι πολύ μικρές. <coughs> Αναμένουμε λοιπόν από τον πατέρα που θέλετε να είστε να ορίσει σωστά τις προτεραιότητες γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο παιδί χρειάζεται περισσότερη ενθάρρυνση από τα άλλα για την ώρα. Το είπα αυτό προηγουμένω ε, με χαμόγελο βέβαια. Δεν θέλω να μονοπολίσω το δικαίωμα της πατρότητας. Ε, όλοι καλείστε να αναλάβετε το ρόλο του πατέρα ή της μητέρας. Γνωρίζουμε πως η επιτυχία έχει πολλούς γεννήτορες, ε, αλλά νομίζω πως όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους. Όσο περισσότερο τα καταφέρνουμε, όσο καλύτερα τα καταφέρνουμε ε, και να παρουσιάσουμε τον αντίκτυπο της περιφερειακής πολιτικής και ήταν μάλιστα καιρός ε, να δημιουργηθεί μια μονάδα που θα ασχολείται με την αξιολόγηση τόσο περισσότερο λοιπόν θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ε, οι συνθήκες σε πλαίσιο, οι δημοσιονομικές ε, θα ε, ακολουθούν. Είναι δύσκολο πριν από την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προπολογισμού να προβεί κανεί σε οποιαδήποτε δήλωση. Θα μπορούσα απλά να πω ότι η τάξη μεγέθου σε ποσοστά είναι μια κατεύθυνση, ένας προσανατολισμός που θα χρησιμεύσει ε, ως μέτρο. Τώρα, πότε ακριβώς θα φτάσουμε σε αυτό δεν ξέρω. Η συνέχεια των ακροάσεων θα το δείξει. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά θα χρειαστεί και η στήριξή σας για να επιτύχουμε. Διότι δεν μπορούμε να πούμε, όπως λένε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο τάδε επίτροπος είναι που έχει το μεγαλύτερο προπολογισμό, το, το, το, δεύτερο μεγαλύτερο κτλ. Αυτό δεν είναι σημαντικό για μένα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όλοι οι θύνοντες να κατανοήσουν ότι μόνο με μια προσέγγιση περιφερειακής συνοχής θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη της Ευρώπης στις περιφέρειες και εάν μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε, αν μπορέσουν να το καταλάβουν οι περισσότεροι ώστε οι σκέψεις που σας ανέφερα προηγουμένως ότι δηλαδή και άλλες πολιτικά οράματα μπορούν να, να υπάρχουν, τόσο περισσότερο θα τα καταφέρουμε να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους. Εγώ πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Κυρία Κάντενμπαχ, δύο πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Μιλήσαμε σήμερα για την καλή συνεργασία, για ένα θέμα συνεργασίας με τις πόλεις. Ε, μπορούμε να αναμένουμε ε, ε, και κανονισμό σε θέματα εταιρικής σχέσης. Η Πρόεδρος. Ε, χαιρετίζω τον κύριο Λούκη Φαντεμπράντεν που βλέπω εδώ το, ε, μεταξύ μας. Θα είμαστε ε, ευτυχείς να συνεργαστούμε μαζί σας με την Επιτροπή των Περιφερειών δηλαδή, η οποία ενισχύθηκε με την συνθήκη, επέκτησε περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητες. Είμαι πεπισμένος ότι ο Λούκο και η ομάδα του θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτές τις επιπλέον. Οι περιφέρειες έχουν 350 εκπροσώπους στην Επιτροπή των Περιφερειών. Αποτελούν λοιπόν μια πηγή εμπειρία στην οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ε, εταιρικής σχέσης, ε, ειλικρινά θα πρέπει να ασχοληθώ με το θέμα. Ε, αν αυτό είναι χρήσιμο και σκόπιμο, θα ξεκινήσω την, την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Ο Πέτρου Κωνσταντίν Λούχαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε για τις ε, σαφείς σας αυτές τις απαντήσεις. Το να απολοποιηθούν οι κανόνες είναι μια αναγκαιότητα στο πλαίσιο της ε, ε, της κινητοποίησης των προγραμμάτων και της καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. Το πρώτο πακέτο των μέτρων απλοποίησης έχει οθετηθεί το περασμένο Απρίλιο και ήδη τίθεται σε εφαρμογή και ένα νέο πακέτο ελπίζουμε πως θα ξεκινήσει πολύ σύντομα λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των σημαντική για χρήση των διευθυντικών ταμείων ε, με τη μέγιστη αποδοτικότητα προβλέπετε νέα πλουστευτικά μέτρα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και πώς σκέφτεστε να βρείτε μια ανισορροπία ανάμεσα στην απλοποίηση και τον έλεγχο που είναι σίγουρα απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ε, Letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage, <laughs> aushalten ist immer ein Problem. Aber Πάντοτε είναι δύσκολο κανείς να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις και απαιτήσει. Έχετε δίκιο σε σχέση με, το, με την τρίτη δέσμη, την απλουστευτική. Τώρα περνά στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ληφθεί μια σχετική απόφαση. Οπότε θα εξετάσετε το κείμενο και θα δούμε πώς θα πάμε. Και νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν επιδείξει ευελιξία, τόσο ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε τις αναγκαίες αλλαγές. Πάντω, υπάρχουν και κάποια όρια σε όλε τι προσπάθειες, σε όλε τι δυνατότητε. Ίσως κανείς θα πρέπει να περιμένει, να δει στην πράξη τι γίνεται, διότι και οι τρεις προσπάθειες ε, απλούστευσης αποσκοπούσαν στο να γίνουν τα πράγματα απλούστερα. Να δούμε επομένως πώς θα πάνε τα πράγματα να δούμε. Τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε φυσικά να φημώσουμε κανέναν. Ε, αυτούς εκείνοι, δηλαδή οι οποίοι σκέπτονται ότι θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω μεταβολές. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Επομένως, γιατί να μην κάθε κανείς να σκέφτεται τι μπορεί να γίνει περαιτέρω στο μέλλον, όμως το πιο βασικό είναι να δούμε κατά πόσο τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν υιοθετηθεί κατά πόσον πετυχαίνουν τους τεθέντες στόχους. Επομένως, εάν τελικά προκύψει ότι το σύστημα είναι στέρεο, σταθερό, τότε θα κάτσουμε να σκεφτούμε τι περαιτέρω μπορούμε να πετύχουμε. Κύριε υποψήφιο, ε, έχω ήδη υποβάλει κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένα. για τους ισχυρισμούς εκείνους ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει αποφανθεί για την περιφερειακή πολιτική και την διαχείρισή της. Εσείς, τι θα κάνετε, θα συμφωνήσετε για την συνδιαχείριση αυτήν ή θεωρείτε ότι η συνδιαχείριση εγκυμονεί κινδύνους, δεύτερον και συγκεκριμένο. Περιμένουμε και άλλες εκθέσεις σχετικά με την πολιτική συνοχή όμως, επί τη βάση των όσων σήμερα γνωρίζουμε. Θα συμφωνούσατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν οι στόχοι 1, 2 και 3. Και κάτι άλλο τώρα που είναι πιο πολιτικό ζήτημα. Εσείς προτίθεστε μαζί με εμά την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής να αναζητήσουμε περισσότερα κονδύλια για την περιφερειακή πολιτική. Also, wir können die Regionalpolitik δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει περισσότερο παραπέρα η περιφερειακή πολιτική εκτός εάν υπάρχει ε, ένα τέτοιο μοντέλο συνδιαχείρισης. Θα προσπαθήσω εγώ πάντως να ελοπίσω τους στόχους μας και ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατόν να γίνουν όλοι οι σχετικοί έλεγχοι. Οπότε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε σε θέματα ουσίας. Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου στις χώρες μέλη και αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντως αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας. Αυτός είναι ο στόχος που θα παλέψουμε να πετύχουμε και αυτό θα το μελετήσουμε κατά την θητεία μου όπως κάναμε και στο παρελθόν. Στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να κάτσουμε και να εξετάσουμε κατά πόσον πέραν των ετησίων εκθέσεων θα πρέπει να έχουμε δηλώσεις ε, και θέσεις πιο αποφασιστικές από τα κρατημέλη όσον αφορά τους ελέγχους για τον τρόπο διαχείρισης των οικοδηλίων Ήδη εθελοντικά το έχουν κάνει αυτό κάποια κρατημέλη. Θα πρέπει όμως και οι 23 τώρα να προσπαθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, ε, είμαστε προσιλωμένοι στους στόχους μας. Και επομένως, να θεωρήσουμε ότι η περιφερειακή πολιτική καλύπτει όλα. Η δε συνεργασία θα πρέπει να είναι ζήτημα τη σημασία στο μέλλον και προτεραιότητα. Ήδη έχουμε εξαντλήσει, έχουμε ζητήσει πάρα πολύ το θέμα του προπολογισμού. πάντοτε Υπουργείο Οικονομικών λένε δεν έχουμε, υπάρχουν αρκετά λεφτά. Εμεί όμω πάντοτε με τη σειρά μα μπορούμε να δίνουμε τη μάχη μα. Να ζητούμε περισσότερα. Θα πρέπει επομένω να έχουμε κάποια επιχειρήματα και να προσπαθούμε να αποδείξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τη ε, περιφερειακή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι για την πειθαρχία αλλά και την αποτελεσματικότητα. Το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο ε, το έχουμε επιστατεύσει ε, εδώ και χρόνια πολλά για ε, τα προγράμματα που θα φτάνουν μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 9 και υπήρξε παράταση. 3% των των, των πιστώσεων. 2,5-22% από τα κράτη-μέλη όμως ήταν κάτω από το μέσο όρο όσο αφορά την εκτέλεση. Και 370% είναι η διαφορά του καλύτερου από τον χειρότερο για το ένα ταμείο. Οπότε έχουμε 45 δις τα οποία τελικά δεν απορροφήθηκαν, χάθηκαν. Να δούμε τι θα γίνει με το Μισογείο στο τέλο τη χρονιά αυτή. Για πετε μα εσεί, πώ βλέπετε το ρόλο σα. Θα κάνετε κάτι για να υπάρχει καλύτερη απορρόφηση των πόρων. Προτίθεστε να έχετε κάποια μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και περισσότερη διαφάνεια. Όχι άλλη διπλωματία. Να κατονομάζετε τις χώρες και να λέτε ε, ότι υπάρχουν διαφορές και γιατί υπάρχουν αυτές τις διαφορές. Ούτε το 2013 έχουμε καλέ επιδόσει. 300% είναι διαφορά μεταξύ των καλών μαθητών και των κακών μαθητών. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξετε τα πράγματα. Es Επίτροπος. Είναι θέμα της capacity building, είναι ένα γενικότερο θέμα. Άρα θα πρέπει να έχουμε περισσότερο capacity building στο μέλλον και το ξέρουμε. Και να δούμε ποιες χώρες δεν μπορούν να εκτελέσουν τα προγράμματα μέσα στις τεθήσεις προθεσμίες και μπορούν ή δεν μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια. χρειάζεται capacity building, δημιουργία δυνατότητών γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητε φαίνεται ή και δεν υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη. Ε, χρειάζεται κατάρτιση, εκπαίδευση, ε, όπου χρειάζεται να γίνεται. Τώρα ρίχνω μια ματιά στι πιο πρόσφατε εξελίξει. Τι έγινε πέρσι. Πέρσι καλύφθηκε πάρα πολύ το χαμένο έδαφο όμω. Υπήρχαν προβλήματα με την εκτέλεση. Λόγω της ε, οικονομικής κρίσης. Οπότε κάποιες εταιρείε οι οποίες ε, θα έπρεπε να συμμετέχουν ανησύχησαν πάρα πολύ με το πόσο άσχημα πήγαινε η συγχρηματοδότηση. Ελπίζω επομένως ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει και το οφείλεται απλώς στην δυσμενή συγκυρία. Έχουμε και άλλες δυσκολίες διαφορετικό χαρακτήρα. Βέβαια, είναι περίπλοκες και οι νομικές διατάξεις που διέπουν αυτή την πολιτική. Υπήρχαν προβλήματα ευθύ εξ αρχή την περίοδο 2000-2006. να κοιτάξει και να αναλύσει καλύτερα τα αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχει κάτι σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα και κάτι λέει ένας καθηγητής όπου πρότεινε ότι έχουμε πάρα πολύ σταδιακά φτωχά αποτελέσματα από τα κρατημέλη. Τις τελευταίες 27 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε πάνω από τέσσερα δις για το περιφρακό και το κοινωνικό ταμείο. 30 και 57% δηλαδή αύξηση σε σχέση με το κάθε ταμείο. Δηλαδή, επομένω, τι έλεγχο είναι αυτό, τι, τι, τι, τι, τι ποιοτική πολιτική να γίνει. Αφού κατά αυτόν τον τρόπο εκταμείωθηκαν τα χρήματα, είναι αυτές οι προτάσεις Μπάρκερ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Χρειάζεται η μια πειθαρχία. Ωραία, έχουμε κάποιε εκθέσει τη Γενική Διεύθυνση τη περιφερειακή πολιτική. Αλλά δεν έχουμε καμία σοβαρή εκθέση από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη θα υποβούν κάποιε εκθέσει που θα αποτιμηθούν. Και στρατηγικέ εκθέσει. για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Και αυτό θα καλύψει και την ε, οικονομική πτυχή, αλλά και την ουσία. Οπότε, και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε που βρισκόμαστε στη συνέχεια, δε, θα πρέπει να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη στην επόμενη περίοδο, στο επόμενο πρόγραμμα. Άρα, να κάτσουμε για να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση του που βρισκόμαστε και να δούμε τι χρειάζεται να αλλάξει. Βόιτσεχ Ολέινιτσαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δεν έχουμε μισά ζητημάτων. Πρώτα πρώτα είναι οι στόχοι. Βάλατε κάποιους νέους στόχους για την πολιτική της συνοχής. Ανάπτυξη, παιδεία, θέσεις απασχόλησης όμως Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις παραδοσιακές προσπάθειες ούτως ώστε κάτι να γίνει με, τα, με την υποδομή, ιδίω στα νέα κράτη-μέλη, γιατί εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Από πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα. Δεν πρόκειται να έχουμε αύξηση του προπολισμού μετά το 2013 γιατί αυτό προβλέπει η πολιτική που έχει χαρακτή. Άρα, εσείς τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε για την Ήπεθρο. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο προγράμματα για την Ήπεθρο. Πρώτα-πρώτα είναι τα προγράμματα της ε, πολιτικής συνοχής αλλά και της ανάπτυξης της Ήπεθρο. Επομένως, πέστε μου την προσωπική σας άποψη Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μία και μόνη πολιτική για τις ε, περιοχές στην Ήπεθρο. Αυτό το οποίο αναφέρεται ήδη καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε προγράμματα και έργα υποδομής, εκεί που χρειάζονται. Ήδη θα προβλέπονται από το Ταμείο Συνοχής και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Α, τι, λέγαμε, μισό λεπτό, έχασα τη σειρά. Α, ναι, ναι, λέγαμε για, το, για την Ήπεθρο και τους Ευρωπαίους που ζουν στην Ήπεθρο. Ναι, αξίζει της προσοχής μας, γιατί προβλέπονται και οι πόροι που χρειάζονται. Δεν θα τον μπερδεύουμε πολύ όσον αφορά την κατανομή των πόρων και το τι θα γίνει με τα ταμεία. Θα πρέπει να δούμε πού σκοπούν όλα αυτά, ποιος είναι ο τελικός στόχος. να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο κάθε προγράμματο και να δούμε πού χρειάζεται να κάνουμε κάποιο είδου εναρμόνιση, κάποιο είδου ε, προσαρμογή των προγραμμάτων, ώστε οι τελικοί χρήστε να ωφελούνται και να γίνουν ζωή του πιο εύκολη. Θα πρέπει να αποφύγουμε τι επικαλύψει. και θα πρέπει ομένω οι ενισχύσεις να μην επικαλύπτονται αλλά να έχουν σωρευτικά θετικά αποτελέσματα. Ε, you already mentioned your support for programs which integrate. Ε, Είπατε ήδη ότι θα βοηθήσετε τα προγράμματα, τα περιφερειακά ε, όπου χρειάζεται, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω τι προσέγγιση υιοθετείτε όσον αφορά κάποια προγράμματα πόλη περιφερειακά που αφορούν κάποια συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόβλημα ε, ανάπτυξη στην Ανατολική Πολωνία και αυτό το πρόγραμμα ε, συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο και θα αρχίσει να τρέχει το, άρχισε να τρέχει το 2007. Θεωρείται ότι τέτοιου είδου ε, πολυπεριφερειακά προγράμματα είναι κάτι το χρήσιμο, τόσο ώστε να λυπηλήσουμε κάποια προβλήματα, προβλήματα υπανάπτυξης σε κάποιες περιφέρειες. Θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να συνεχιστούν και κατά την επόμενη ε, χρήση, επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Δεν έχω επερώτηση, οπότε σας ε, ρωτώ τώρα το εξής. Αυτά τα προγράμματα τα πολύ περίεργα, πώς τα βλέπετε. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πολύ συχνά αξιολογούνται πριν αποδώσουν κάποιους καρπούς πριν δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσει κανείς τι θα τα κάνει ε, πολύ νωρί. πριν βγάλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μήπως θα έπρεπε να τρέξουν επί περισσότερο χρόνο και όχι μόνο επί μία πενταετία. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές όντως θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει υπερπεριφερειακή συνεργασία και αυτό θα πρέπει να γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιληθούν ε, μόνο σε μια περιφέρεια. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερες περιφέρειες για να τα λύσουν. Γι' αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό να έχουμε συνεργασία περισσότερων περιφερειών. Άρα και στο μέλλον θα πρέπει αυτό το μοντέλο να συνεχίσει να ισχύει. Δεν υπάρχει άλλη λύση πολλές φορές. Αυτή η υπερπεριφερειακή συνεργασία πρόκειται για μια τρομερή προσθέμενη αξία για την περιφερειακή πολιτική. Πολλές φορές μιλάμε για την διάρκεια, η παράταση διάρκειας αυτών των προγραμμάτων αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι 7 χρόνια δεν είναι και ε, λίγα, ούτω ώστε να μπορέσει κανείς να τρέξει πρόγραμμα, αλλά και να το αξιολογήσει. Πάντως, γενικά, ε, θεωρώ ακριβώς αυτό, ότι 7 χρόνια είναι κάτι το λογικό. Κύριε Χάν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα του κλιματικού χάους. Στις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο δεν αναφέρεστε καθόλου στα θέματα περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Εδώ εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρξουν εκτός από του κεντρικούς και περιφερειακοί στόχοι. Δεν παίζουν ρόλο τα θέματα αυτά κατά τη γνώμη σας στην πολιτική συνοχής. Και επιπλέον, τι σχεδιάζετε να κάνετε απέναντι στη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κλιματικούς στόχους μέσα από τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Έχετε μιλήσει για διαφάνεια. Με ποιο τρόπο στοχεύετε να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική, διαφανή και στοχευμένη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής από τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τα κονδύλια για το περιβάλλον. Και τέλος, τι σκοπεύετε να κάνετε για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και την ελαχιστοποίηση των λαθών από τα κράτη-μέλη που οδηγούν στη μη απορρόφηση. Ευχαριστώ. Zum Ersten, das ganze Thema Umwelt, Klimawandel, erneuerbare Energie κάθε υπόθεση που αφορά το περιβάλλον, τις κλιματικές αλλαγές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κεντρικά, κεντρικό ζήτημα αυτής της στρατηγικής του 2020 και το είπα στην αρχή ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για τα πιο κρίσιμα σημεία θα πρέπει να αγωνιστούμε η πόλη σας, πούμε, θα είναι ένα από τα κεντρικά σημεία για μένα. Γιατί οι πόλεις είναι αυτές που σπαταλούν ενέργεια. Και ακριβώ με αυτή τη βάση και έχοντας ε, υπόψη μας μια γενική στρατηγική, οφείλουμε να θίξουμε και αυτό το θέμα. Τώρα, εάν σκεφτούμε την ε, δαπάνη των κονδυλίων, θα δούμε ότι πρόκειται για 150 εκατομμύρια ευρώ που πάνε στο περιβάλλον και το κλίμα. Ε, πρόκειται για συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία ε, θα δαπανηθούν κατά τη διάρκεια αυτή της προγραμματική περίοδου. Πολλά έχουν συμβεί. Υπάρχει το πακέτο της απλοποίηση και Αυτό σε σχέση με τις ε, κατοικίες, στον τομέα μάλλον των κατοικιών, μπορούμε να αυξήσουμε την ε, ενεργειακή επάρκεια και αποδοτικότητα. Ήδη έχουν γίνει πολλά. Και θα μπορέσουμε να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις εργασίες. Στα κράτη-μέλη υπάρχει μια γενική εικόνα για το ποιο είναι ο δικαιούχος κάθε προγράμματο, Η παρουσίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι εναρμονισμένη. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές παρουσίαση, πράγμα το οποίο ε, οδηγεί σε επικρίσεις και αυτό θα είναι ένα σημείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί την επόμενη περίοδο. Θα μιλήσουμε δηλαδή και για αυτό το θέμα. Και έπειτα η αρχή της ε, επικουρικότητας ε, εδώ ισχύει. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να γίνει και αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρόεδρος, νομίζω πως μπορούμε να μείνουμε σε αυτό τους ε, κανόνες. Ε, είναι πιο αισιόδοξη η κατάσταση με το ρολόι αυτό. Θα έχουμε ακόμα μια ερώτηση. Ο κύριος Βλάσα αντικαθιστά τον κύριο Κούρσκι. Πάει πίσω. Ναι. Ο Παύλο Αμέσχη στο έγγραφο προσανατολισμό αναφέρθηκε στην πιθανή μεταφορά του της ποιότητα ζωής και της διαφοροποίησης της οικονομίας καθώς και της πρόσβασης για την ε, μετακίνηση κονδυλίων από την κοινή γεωργική πολιτική στην ε, πολιτική συνοχή. Ξέρω από τις συζητήσεις ε, στην Επιτροπή Περιφερειών με δημάρχους ή τοπικούς ηθήνοντες ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο λόγω των τρεχουσών δυσκολιών. Εσείς τι πιστεύετε είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο. Ναι, ξέρω το έγγραφο, ξέρω το έχω διαβάσει. Ξέρετε ότι την ενεργική πολιτική εγώ θα ήθελα να την αφιερώσω σε άλλα πράγματα και όχι σε θέματα ανταγωνισμού. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο, αλλά αυτό που είναι καθοριστική σημασία είναι να είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε τα δύο προγράμματα. Οι επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί και που είναι αιτιολογημένες ε, λένε πως υπάρχει, γίνεται ομοδοποίηση των δύο προγραμμάτων και αυτές τις κριτικές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και πιτα το ποιος θα είναι αρμόδιος για μένα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Έχουμε μαζί μας τον Λουκ Βαντεμπράντεν και θα μείνουμε πιστοί στην παράδοσή μας και θα δώσουμε ένα λεπτό ή ενάμιση λεπτό ε, στον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών. Έχει το λόγο, Λουκ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή μου πρόεδρε, αγαπητή Ντανούτα. Αγαπητέ υποψήφι επίτροπε, το μέλλον της πολιτικής συνοχής είναι ένα θέμα που, είναι, που, που μάλλον αφορά την γενική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θέμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την εφαρμογή των διαφόρων στόχων όπως η στρατηγική του 2020, είναι μια πολιτική που στόχο έχει να συμβάλλει στις ε, διαφορές ευκαιρίες ανάπτυξης που έχουν οι περιφερειές μας και έτσι να μπορέσει να προσαρμοστεί στις διάφορες ε, περιφέρειες και καταστάσεις μέσα στο πλαίσιο ε, των διαφόρων ε, περιφερειών. Με στόχο λοιπόν της ένταξης ε, της περιφερειακής συνοχής στη συνθήκη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο εδαφικός αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός. Όλες οι περιοχές θα πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό, ότι έχουν δηλαδή εδαφικό αντίκτυπο οι δραστηριότητές τους και να γνωρίζουν τον αντίκτυπο αυτών. Φτάσαμε σε ένα τελικό ορισμό της ε, δαφικής ε, συνοχής και ξέρετε αγαπητή Πρόεδρε ότι ε, εμείς λέμε πως θα πρέπει να συμπληρώσουμε τις ελευθερίες που ήδη θεσπίζονται από τη συνθήκη μέσω της προσθήκης των, της επιπλέον ελευθερίας των πολιτών να μπορούν να επιλέξουν πού θα ζήσουν και πού θα εργαστούν παρά τις, τα υπάρχοντα γεωγραφικά ζητήματα που θα μετατρέψουν σε ουσία ε, ανταγωνιστικότητα σε αυτά που στιγμής θεωρούνταν εδαφικό μειονέκτημα. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές να λάβουν υπόψη τους στόχους της εδαφικής συνοχής στο σχεδιασμό της εφαρμογής και της αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, να αποφύγουμε τον, την τομεοποίηση και ελπίζουμε πως θα εξασφαλίσετε αυτό, αυ, αυτές τις προσδοκίες. Επίσης, μιλάμε για απομάκρυνση από την πιο επιτυχημένη, ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης ε, εναντί όλων των μορφών επανεθνικοποίησης. Ε, η πολιτική συνοχή έχει αποδειχτεί εξαιρετική στρατηγική που, έχει, που επιτυγχάνει δύο στόχους, να εφαρμόσει δηλαδή τους κοινοτικούς στόχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και άλλο στόχος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και περιφέρειες να επιτύχουν από κοινού τους στόχους τους. Τέλος, παρακαλώ η Επιτροπή, πιστέψτε περισσότερο από ό,τι παλιότερα στην πραγματική σημασία της πολυεπίπεδης κυβέρνηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε και όχι απλά να λέμε ότι είναι ένα είδος θεωρητικής προσέγγισης. Χρειάζεται να υπάρχει. Και επιτά, έχω την εντύπωση πως ε, μιλάτε πολύ σχετικά με τις περιφέρειες και τις πόλεις θα πρέπει όμως να μπορέσετε να συνομιλήσετε άμεσα με τις πόλεις και τις περιφέρειες ως πραγματικούς εταίρους. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πιστεύω λοιπόν και είμαι πεπισμένος ότι όταν δώσω κάποια στοιχεία του πιστεύω της Επιτροπής των Περιφερειών ότι φυσικά δεν είστε μόνο ευπρόσδεκτο. δεν χρειάζεται να σας πω ότι είστε ευπρόσδεκτο στην επόμενή μα Ολομέλεια το Φεβρουάριο, αλλά είμαι βέβαιος ότι και πρώτα απ' όλα με τους τοπικούς και περιφερειακού ηθήνοντε άμεσα θα συνεργαστείτε για να επιτύχετε. Και αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, αλλά και εσείς ως κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης. Να ενεργήσουμε όλοι από κοινού με μια πραγματική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Η ακρόαση φτάνει στο τέλος της. Επισήμως, αν ο ψήφος επίτροπος θέλει οπωσδήποτε να πει δύο λόγια, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια αυτού του απογεύματο ε, πέρασα διάφορους, από διάφορους ρόλους, από πατέρας ε, σε άτομο μηχανή, ε, κινητήριος δύναμη. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το μεγάλο σας ε, ενθουσιασμό. Μου δίνει αυτό μια ιδέα για το τι με περιμένει, αλλά και το τι σας ενδιαφέρει και τι σας ανησυχεί και θα πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι αν είχαμε τη δυνατότητα θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να συνεργαστώ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών μαζί σας και βεβαίω θα κάνω λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος, δεν είναι λάνθαστος, αλλά μπορώ να πω και αντίστροφος ότι και ίσως μάλιστα τολμώ να πω ότι εσείς δική εσείς θα ψηφίσετε υπέρ κατά των όσων σας προτείνω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα των περιφερειών, θα αγωνιστώ για τις περιφέρειες και φυσικά θα επισκεφθώ τις περιφέρειες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έχω το ίδιο πρόγραμμα τόσο φιλόδοξο όσον αφορά τις μετακινήσεις της κυρίας Κιούμπινερ αλλά είναι σαφές ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει τι συμβαίνει επί τόπου για να μπορεί μετά να συζητήσει γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ έντιμη, ειλικρινή και επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Please, colleagues, don't, don't... Συνάδελφοι, παρακαλώ μην φύγετε από την αίθουσα γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε για το τι θα κάνουμε. Καταρχήν ε, θα ήθελα επισήμως να ευχαριστήσω, σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ κατά τη διάρκεια των τριών ωρών και τον υποψήφιο επίτροπο που επιβίωσε. Ο Μάρκ Τουέν είπε κάποτε ότι το χειρότερο είδος ε, θανάτου είναι το να μιλά κανείς μέχρι θανάτου, αλλά πιστεύω πως αυτό το ξεπεράσαμε ε, αυτές τις τρεις ώρες καρποφόρων ε, ανταλλαγών απόψεων. Τώρα θα κάνουμε μισή ώρα διάλειμμα και στις 8 θα συναντηθούμε όλοι και πάλι για την αξιολόγηση. Εννοώ όλους τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων ε, που θα συνοδεύονται από τους ε, βοηθούς τους και τα μέλη της γραμματείας θα είναι μαζί μας. Παρακαλώ λοιπόν χρησιμοποιήστε αυτό το μισάωρο, ελάτε σε επαφή με τις ομάδες σας και αποφασίστε για την αξιολόγησή σας. Και στις 8 θα τα πούμε στην αίθουσα Α1G3. Να είστε στην ώρα σας λοιπόν στην αίθουσα παρακαλώ. Ευχαριστώ.